Okay, good afternoon. Καλησπέρα σας. Ένα θερμό καλώς όρισμα. Θερμό τονίζω, καθώς καριζέστηκε μέσα και έξω από το κτίριο. Χαίρομαστε που σας βλέπουμε εδώ στην, ε, στο διάλογο του άρθρου 17. Μια πολύ σημαντική πλατφόρμα για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα. Θα συζητήσουμε εδώ το ρόλο των εκκλησιών και των θρησκειών για την εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα. Ε, οι δερμηνείς σας ενημερώνουν ότι βρισκόμαστε στην 22η ημέρα των κινητοποιήσεων που κάνουμε και ακόμα δεν έχουμε δει καμία αντίδραση εκ μέρους της διοίκησης. Αντίθετα, ο Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σκληραίνει ακόμα περισσότερο τη στάση του. Στη σημερινή συνεδρίαση, πολλοί συναδελφοί μα έχουν επιταχθεί και είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν. Σε ένδειξη αλληλεγγύη, η ελληνική καμπίνα δεν θα προχωρήσει σε στάση εργασία όπω αρχικά προβλεπόταν. Ωστόσο, η διερμηνία θα διακοπεί ακριβώ στην προγραμματισμένη ώρα λήξη τη συνεδρίαση. Και συνεχίζουμε με την κυρία Μαγκίνες. Θα έρθει ο κύριος ε, Ταγιάννη αργότερα για να συμμετάσχει στο διάλογο. Εδώ έχω τον κύριο Τζάιε, βλέπετε όσο πιο συχνά το επαναλαμβάνω το όνομα τόσο πιο λάθος το προφέρω, αλλά θα σας αποκαλώ Λούκα μια και γνωριζόμαστε τόσο καλά. Πριν λάβετε τον ε, τίτλο του Προέδρου ε, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ήταν ήδη πολύ γνωστός. Ε, εμείς από παραμεθόριο περιοχή της Ιρλανδίας που, αφορά ιδιαίτερα το Brexit, σας γνωρίζουμε πολύ καλά, σας γνωρίζουν οι πολίτες, σας γνωρίζουν όλοι. Ε, Λουκάι, αν δεν έχεις αντίρρηση, μπορείς να με φωνάζεις Μουρέιτ. Πάντως, ως πρόεδρος έχει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη συζήτησή μας. Τους τελευταίους 18 μήνες ε, του διαλόγου ακούσαμε με ικανοποίηση διάφορες ε, προτάσεις για την εικόνα τη γενικότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μέλλον της, συζητήσαμε θέματα ανάπτυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ελευθερίας ε, θρησκευτική, ε, ελευθερίας θρησκευτικής πεπιθήσεως και έτσι έχουμε τώρα σταθεί στο θέμα των ε, κοινωνικών δικαιωμάτων ως κομμάτι της εσωτερικής πολιτικής. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εσείς τι έχετε αποκομίσει, τι βλέπετε ότι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά ενδεχομένω που έχουμε επιτύχει συγκεκριμένους τομείς πολιτικής αναζητώ, εκεί που μπορούμε να αναπτύξουμε δραστηριότητα και πέραν των όσων κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα λοιπόν τις δικές σας προτάσεις. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνω ότι έχουμε και δύο επιφανείς τρελέχοι της Επιτροπής ε, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περίνσκη και Ζάμπον, που θα αναλάβουν την ε, καθοδήγηση των εργασιών μας, τα δύο πάνελ που έχουν προβλεφθεί και η συμπερίληψη και ε, χώρος εργασίας είναι οι δύο τομείς μας. Οι αποφάσεις του Προεδρείου ε, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον κοινωνικό διάλογο ε, και τη συνεργασία με μέσω και των αντιπροσωπιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν αυτό να το διερευνήσουμε περαιτέρω, να εξασφαλίσουμε στο δυνατόν πιο αποτελεσματικό διάλογο για όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό και πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Γνωρίζω ότι η τωρινή μορφή συνομιλιών που έχουμε έχει τα ωριά της, αλλά θα ήταν καλό να κοιτάξουμε περισσότερο την αποτελεσματικότητα των εκδηλώσεών μας και βεβαίως γι' αυτό σας παρακαλώ να μου πείτε αν βλέπετε κάποιο τρόπο βελτίωσης της μεθοδολογίας μας. Ο στόχος του διαλόγου είναι να, να χτίσουμε πάνω στη βάση αυτή τα σοβαρά θέματα της κοινωνικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει πολύ ενέργεια για να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας και θεωρούμε ότι έχει δοθεί υπερβολικά πολύ έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και τα στατιστικά κυρίως στοιχεία ως ορόσημα της ε, προόδου, χωρίς όμως να εξετάζουμε εάν είναι ισο, ίση και ισότιμη η κατανομή των ωφελημάτων αυτής της οικονομικής ανάπτυξης. Ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων στον Γκέτεμπορκ αποτελεί μια απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολλά τα κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και γι' αυτό χρειάζεται οργανωμένη και συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο και γι' αυτό και η χρηματοδότηση και γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε όλα τα προγράμματα και αυτά των οποίων η χρηματοδότηση είναι υπό το, την αιγύδα των κρατών μελών. Βεβαίως έχουμε πάνω απ' όλα το χάρτη των θεμελιωδών ελευθεριών και των δικαιωμάτων. Είδαμε πόσο δύσκολες συνθήκες αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λιγότερο κινητικοί, γιατί θεωρούνται παράγοντες παραγωγής σε μια αγορά εργασίας. Θα το συστήσουμε και αυτό οι, αγο... οι θρησκείες, οι εκκλησίες, οι θρησκευτικέ οργανώσεις μπορούν να συμβάλλουν στη συζήτηση αυτή. Πολλές είναι οι εκκλησίες που εκπροσωπούνται εδώ και που ε, δραστηριοποιούνται στην, ε, στο να υπογραμμίζουν τη σημασία της ανθρώπινης διάστασης του κοινωνικού αυτού πυλώνα. Ξέρω ότι πολλοί από εσά είχατε άλλωστε και συμμετοχή στη Σύνοδο του Γκότεμπουργκ. Ωστόσο, και σε νομικό επίπεδο ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να προωθήσουμε τους νόμους που θα πρέπει να υιοθετηθούν σε μακροεπίπεδο δηλαδή. Σε μικροεπίπεδο πρέπει ο καθένας να αναλαμβάνει και τις ευθύνες του στα όσα συμβαίνουν καθημερινά, μέρα με τη μέρα. Για το σημερινό σεμινάριο η Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει κάνει μελέτες και έχετε το κείμενό τους, την έκθεσή τους ε, στο φάκελό σας δείχνει ότι χρειάζεται και η συνεργασία, η συμβολή των εκκλησιών και θρησκευτικών οργανώσεων, καθώς είναι παρούσες στις τοπικές κοινωνίες πάντα. Έχουν εκπροσώπηση επίσης στις Βρυξέλλες, μπορούν να συμβάλλουν στην ε, διαμόρφωση στρατηγικών επιλογών. Ταυτόχρονα είναι παρούσες ε, στη ζώσα κοινωνία σε τοπικό επίπεδο. Η συνεργασία λοιπόν με τις εκκλησίες και τις θρησκευτικές οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να δώσει πολύ σημαντικά στοιχεία προς, την, προς τον κοινωνικό διάλογο και την πρόοδο. Βεβαίως κάθε κράτος έχει τις ιδιαιτερότητές του και βέβαια τις ε, ιστορικές καταβολές. Είναι μεγάλη συμβολή των εκκλησιών και των θρησκευτικών οργανώσεων και σε, φιλανθρωπικό, σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες και άλλες. Μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπληρώνει τις ε, προσπάθειες των κρατών μελών χωρίς καμία διάκριση ως προς το αν πρόκειται να στηριχθεί μια θρησκευτική ή μια μη θρησκευτική οργάνωση. Πάντως, ε, ιδιαίτερα τιμούμε τη συμβολή των εταίρων μας από τις θρησκευτικέ κοινότητες και τις εκκλησίες. Σήμερα δίνεται η ευκαιρία να ακουστεί η φωνή σας και ταυτόχρονα να ε, τονιστεί ο ρόλος της κοινωνικής βοήθειας και συνεργασίας που προσφέρεται. Η κοινωνική πρόοδος και η εκκοσμίκευση είναι χωριστές διαδικασίες. Δεν ε, παρεμβαίνει μία στο πεδίο της άλλης. Έχουμε μία πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δημοσιεύθηκε αυτό το μήνα που δείχνει ότι δύο τρίτα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτίζονται με μία θρησκεία ή δηλώνουν ότι ανήκουν σε μία θρησκευτική σε μία εκκλησία. Επομένως μπορούν να βρουν απαντήσεις στα προβλήματά τους χάρη και στη συμβολή των εκκλησιών και των θρησκευτικών οργανώσεων. Ε, σεβασμιότατη αδεσιμότητα, κυρίες και κύριοι, έχω έρθει για να σας ακούσω, όπως πάντα, να μάθω από σας και να μπορέσω να μεταφέρω το μήνυμά σας σε όσους είναι δετεθειμένοι να μας ακούσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άλλα λόγια σήμερα από μένα δεν θα ακούσετε. Ήθελα απλώς να περιγράψω τα δεδομένα μέσα στα οποία θα γίνει η συνεδρίασή μας με χαρά παρακαλώ τον πρόεδρο Λούκα της ΕΟΚΕ να αναλάβει τα ενία. Αισθάνομαι πάντα ότι είμαι ταπεινή μπροστά του και τον παρακαλώ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε Μαρίντ. Ελπίζω να κατάφερα να προφέρω σωστά Ιρλανδικά το όνομά σου. Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ ε, σήμερα μαζί σας και θέλω να χαιρετήσω όλους τους σεβασμιότατους, εδεσιμότατους ευρωβουλευτές καθώς και κάποιους φίλους από ευρωπαϊκές οργανώσεις που βλέπω ότι είναι παρόντες σήμερα και χαίρομαι πολύ που είστε εδώ μαζί μας και εγώ που είμαι μαζί σας. Για πολλούς λόγους. Πρώτον γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία ε, του θεσμικού οργάνου στο οποίο βρισκόμαστε καθώς και του διαλόγου στο πλαίσιο του άρθρου 17. Ε, είναι πραγματικά εξαιρετική αυτή η δυνατότητα που μας δίνει το άρθρο 11 της συνθήκης αν και δυστυχώς θεωρώ ότι δεν έχει εξοποιηθεί πλήρως. νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ακόμα δυνατότητες αξιοποίησης, ακόμα περισσότερες, ε, μεγαλύτερες αξιοποίησης ε, των δυνατότητων που μας προσφέρει το άρθρο 11 ε, και το άρθρο 17. Ακριβώς γιατί καθίσταται δυνατός αυτός ο διάλογος και ελπίζω και στην επόμενη θητεία η Κομισιόν να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση αυτών των δυνατότητων. Ο Πάπας Παύλος ο Έκτος είχε δηλώσει ότι δεν μπορεί να υπάρχει ειρήνη όταν άνθρωποι περιθωριοποιούνται ή αναγκάζονται να ζουν στη φτώχεια. Ξέρετε ότι είμαι καθολικός, ε, για 14 χρόνια παρακολούθησα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ιουσιτών στην Ιταλία και ταυτόχρονα ε, έχω αναλάβει υποχρεώσεις ε, διεθνούς χαρακτήρα στο πλαίσιο της Καθολικής Εκκλησίας. Και αυτή η πολιτιστική και θρησκευτική μου καταγωγή καθοδηγεί και τις σημερινές μου δράσεις. Και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος και με αυτή την ιδιότητα, που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας ε, τόσους διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικές ε, ομάδες και κοινότητες πεπιθήσεων, θρησκείες, εκκλησίες. Γιατί η κοινωνική ε, δικαιοσύνη είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα πνευματικά ζητήματα, τα φιλοσοφικά ζητήματα. Η βοήθεια προς τους φτωχούς και περιθωριοποιημένους ανθρώπους είναι μια κοινή μας αξία όλων των ομολογιών, όλων των ε, κοινοτήτων πεπιθήσεων. Αν δεν υπάρχει αλληλεγγύη, δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή και κατά συνέπεια δεν υπάρχει και κοινωνική ανταγωνιστικότητα, ούτε και βιωσιμότητα, ε, βιώσιμη ανάπτυξη και μέσω της ΕΟΚΕ εγώ είμαι πρόεδρος του θεσμικού οργάνου που εκφράζει την κοινωνία των πολιτών. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η κοινωνική διάσταση αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ένα τρίτο των όσων ε, ε, συναποτελούν τη συνθήκη αφορούν αυτή την κοινωνική διάσταση. Και στο πλαίσιο αυτό η αντιμετώπιση της φτώχειας αποτελεί τμήμα και των ε, στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη που όλο και περισσότερο γίνονται κατευθυντήρια γραμμή για τη χάραξη της πολιτικής μας και για το μέλλον μας. Ταυτόχρονα όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουμε ότι 24% των πολιτών ε, είτε βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας ή απειλούνται από τη φτώχεια. Ε, η νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ε, προβλέπει την ραγδαία μείωση, δραστική μείωση των ανθρώπων που απειλούνται από τη φτώχεια. Η, η οικονομική κρίση δυστυχώ είχε σοβαρότατα πλήγματα σε όλου του Ευρωπαίου, ακόμη και εκείνοι που εργάζονται απειλούνται πολλέ φορέ από τη φτώχεια. Ε, ε, μεγάλα ποσοστά, υψηλότατα ποσοστά ε, ανθρώπων στην Ευρώπη απειλούνται από τη φτώχεια και από την ανεργία. Και αυτό σημαίνει συγκεκριμένα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανάγκη να βελτιώσει την κοινωνική της διάσταση. Η ΕΟΚΕ μαζί και με άλλους φορείς κάνει έκκληση για βελτίωση αυτή τη κοινωνική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γι' αυτό και χαιρετίζουμε θερμότατα τη διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στο Γκέτεμπορκ ω ένα πραγματικά πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Έχουμε συμβάλει πολλάκις και ποικιλοτρόπως στην ανάπτυξη και τη διαμόρφωση αυτής της κοινωνικής διάστασης μέσω της συνεργασίας μας και της εκπροσώπησης των οργανώσεων της ε, κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου χίλιοι ε, εκπρόσωποι ε, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από εργοδοτικές και ε, εργατικές ενώσεις ε, αλλά και άλλες ενώσεις πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχαν πρόσφατα και σε μια σχετική συνδιάσκεψη που διοργανώσαμε η οποία μάλιστα συγκέρασε τις απόψεις ε, που εκφράζει η, ε, η, η κοινωνία των πολιτών όπως είναι για παράδειγμα η προστασία των παιδιών από την φτώχεια που ε, βρίσκεται πλέον ε, κατοχυρωμένη και σε αυτόν τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και αυτό δείχνει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών όταν συνεργάζονται μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής πολιτικής της Ευρώπης. Έχετε επίσης ε, επιλέξει σωστό τίτλο για τη σημερινή μας συνεδρίαση, γιατί η εφαρμογή είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Τα λόγια καλά είναι, αλλά πρέπει να περάσουμε και στη φάση της υλοποίησης και η ΕΟΚΕ εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητεί την κατάρτιση ενό οδικού χάρτη για την εφαρμογή των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να δώσουν κίνητρα, αλλά δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν σχεδόν τίποτα με το 1 ή το 1,3% του ΑΕΠ που βρίσκεται στη διάθεσή του. Επομένω, είναι οι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών και τα κράτη-μέλη, κυρίω σε εθνικό επίπεδο, εκείνοι που καλούνται να εξασφαλίσουν ότι ο ευρωπαϊκό πυλώνα θα εφαρμοστεί στην πράξη και θα σε μετουσιωθεί σε νόμους και σε πρωτοβουλίε, βλέποντα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι η Κομισιόν ε, πρότεινε τη δημιουργία ενό ε, συστήματο βαθμολογία ε, για τα κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Εμεί θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό αυτό, όμω θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει και δυσμευτική επαρκεί αυτή η διαδικασία ακριβώ για να εξασφαλίζεται η καλύτερη υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα. Ταυτόχρονα η Κομισιόν υπέβαλε πρόταση για την ε, θέσπιση μια οδηγία για την εξισορρόπηση τη επαγγελματική και προσωπική ζωή, όπου θα προστατεύονται οι εργαζόμενοι καθώ και υπάρχουν και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προστασία των εργαζομένων και των αυτοπασχολουμένων. Μέσω αυτών των νομοθετικών εργαλείων πράγματι μπορούν να εξασφαλιστούν πολλά. Δεν αρκούν αλλά είναι αναγκαία αυτά. Ε, στις 21 Ιουνίου έγινε το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ ε, και εγώ χαιρετίζω την συμφωνία που αναφέρεται ότι ε, επιτέθηκε σε αυτή, την, σε αυτή τη σύνοδο όσον αφορά την, το συμβιβασμό προσωπικής επαγγελματικής ζωής προστασίας των εργαζομένων. Τα κράτη-μέλη δεν ενέκριναν ακόμη, αλλά οριστικοποίησαν τη γενική τους ε, προσέγγιση προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό ελπίζουμε να ανοίξει το δρόμο για την θέσπιση συγκεκριμένων νομικών εργαλείων πριν από την ολοκλήρωση τη τρέχουσας θητείας και πρέπει πλέον όλοι να καταβάλουν προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρω ότι η Αυστριακή Προεδρία, ε, γιατί συναντήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα με τον ε, Υπουργό Κοινωνικών ε, Υποθέσεων και εργασία ότι υπάρχει η βούληση πλέον να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αυτόν τον κλάδο, σε αυτόν τον τομέα πολιτική. Η απόφαση ΕΠΣΚΟ του Ιουνίου θεωρούμε ότι βαίνει στη σωστή κατεύθυνση και ε, κατέληξε σε μια ισορροπημένη ε, προσέγγιση. Ας δούμε πλέον από εδώ και πέρα ε, αν στη διαπραγμάτευση μπορεί να τεθούν ακόμη πιο φιλόδοξοι στόχοι. Γιατί θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα προσωπικό σχόλιο. Παρατηρούμε ότι υπάρχει και μια τάση να αποδυναμωθεί ορισμένες, ε, ε, ορισμένα στοιχεία ε, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν, για παράδειγμα, την κοινωνική διάσταση των ευρωπαϊκών πολιτικών ή πληρωμένη επαμοιβή γονική άδεια, για παράδειγμα, που μπορεί να ενισχύσει την εξισορρόπηση και την ισοτιμία των δύο φύλων. Ελπίζω λοιπόν όλοι οι συμμετέχοντες στη διαπραγμάτευση να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να ενισχυθεί αυτή η βασική γενική κατεύθυνση της προσπάθειας μέχρι τώρα και όχι να αποδυναμωθεί προκειμένου να καταλήξουμε ε, σε ένα πραγματικά πολύ ε, σημαντικό και θετικό αποτέλεσμα. Αυτό που είπε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Ντόναλτ Τούσκ, να καταλήξουμε σε μια Ευρώπη που θα ε, συμπεριλαμβάνει όλους τους πολίτες και θα νοιάζεται για τους πολίτες της. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε σε κάθε περίπτωση είναι η αδράνεια. Δεν υπάρχει τέτοια επιλογή στο τραπέζι, γιατί αυτό θα ήταν καταστραφικό. Όχι μόνο λόγω της μη υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα, αλλά και διότι κάτι τέτοιο θα απέστελε εσφαλμένο κακό μήνυμα σε όλους τους πολίτες και τους ε, ε, συνομιλητές μας γιατί αυτό θα σήμαινε ότι γυρνάμε την πλάτη στους πολίτες μας και ξέρετε ότι οι πολίτες θα απαντήσουν με τον γνωστό τρόπο διότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι πολίτες δυστυχώς συχνά ε, στρέφονται και κατά των αδυνάμων και κατά των δυνατών Νομίζω ότι μια τέτοια ε, αδράνεια θα, το μόνο που θα μπορούσε να κάνει είναι να ενισχύσει ξενοφοβικές ακρές φωνές και αυτό είναι επικίνδυνο και για την Ευρώπη και για το παγκόσμιο στερέωμα. Η εφαρμογή λοιπόν του κοινωνικού πυλώνα δεν είναι μία από τις πολλές αρμοδιότητες ή απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε, είναι μία από τις βασικότερες απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε και ε, ως ε, επικεφαλής ε, της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη κάνω έκκληση να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα πριν από τη λήξη της θητείας. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας δραστικά για να υλοποιήσουμε αυτόν τον κοινωνικό πυλώνα και να εξασφαλίσουμε και τη χρηματοδότησή του. Έχουμε ήδη ρητός κάνει έκκληση ο κοινωνικός πυλώνας να λαμβάνεται υπόψη στις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο καθώς και στην πολιτική συνοχή. Ε, θυμάμαι τα ξεκάθαρα λόγια του Πρόεδρου Ταγιάννη στο Γκέτεμπορκ όταν είπε ότι πλέον εγκρίναμε τον πυλώνα και πρέπει να δούμε στον επόμενο προπολογισμό να εξασφαλίσουμε και τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτού. Χρειαζόμαστε λοιπόν από τη μία μεριά τα κείμενα, τα νομοθετικά, ταυτόχρονα όμως χρειαζόμαστε σε εθνικό επίπεδο να μετοσιωθούν όλα αυτά τα νομικά κείμενα σε συγκεκριμένε πράξεις και σε χρηματοδότηση. Εμείς καλούμε 30% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να ε, κατευθυνθεί στην ε, διάσταση της ε, κοινωνικής ένταξης και συμπερίληψης ε, μαζί με την παιδεία και την απασχόληση. Άρα πρέπει και αυτή η διάσταση, αυτή η πτυχή της κοινωνικής ένταξης να χρηματοδοτηθεί. Και ε, ε κάτι αντίστοιχο αναφέρεται και ε, σε έγγραφο της Κάριτας Euro που ξέρω ότι συμμετέχει σήμερα στην σημερινή μας συνάντηση. Επίσης, χρειάζονται περισσότερες κοινωνικές επενδύσεις. Είναι αναγκαίες στην Ευρώπη τέτοιες επενδύσεις που θα ενισχύουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις, την κοινωνική επιχειρηματικότητα αυτών των κλάδο της οικονομίας που είναι τόσο σημαντικός και στον οποίο δραστηριοποιούνται πολλές θρησκευτικές και εκκλησιαστικές οργανώσεις που μπορούν πραγματικά να προσφέρουν τη συνδρομή τους στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Αυτό άλλωστε ε, είναι και τμήμα των αποφάσεων που ελήφθησαν τώρα στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου για, μέσω του προγράμματος Investing EU. Και αυτό θεωρώ ότι πηγαίνει στη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω, κυρία Πρόεδρε, και τελειώνω, ότι πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες μας. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή αναγέννηση, αν θέλετε, όπως την αποκαλώ εγώ με ένα συγκεκριμένο μήνυμα για τους πολίτες, με τους πολίτες στο επίκεντρο. Και όπως υπόθηκε και και στις, στους για τα 60 χρόνια από την υπογραφή των συνθήκων της Ρώμης η Ευρώπη βρίσκει την ελπίδα της όταν θέτει στο επίκεντρο των πολιτικών της τον άνθρωπο και αυτό ε, ελπίζω να γίνει το σύνθημα που θα μας καθοδηγεί για το καλό των πολιτών, των λαών, ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να βρούμε τη δύναμη να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες ε, που μας έχουν εναποθέσει οι πολίτες μας προκειμένου να καταστήσουμε δυνατή αυτήν την ευρωπαϊκή αναγέννηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι ήταν εμπνευσμένη η ομιλία σας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω κάποια από τα σκληρά δεδομένα που αναφέρατε. 24% των πολιτών μας απειλούνται από τη φτώχεια. Ακόμη και αυτοί που εργάζονται κινδυνεύουν κατά ποσοστό 1 στους 10-10% από τη φτώχεια. Επομένως τα προβλήματα στον κοινωνικό πυλώνα είναι πολύ βαθιά και πρέπει να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Και βέβαια η υλοποίηση που αναφέρεται έχει κέρια σημασία. Επίσης για τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξέρουμε ότι είναι μεγάλη πρόκληση ο προπολογισμό και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ εύχομαι να συμβεί ένα θαύμα, ίσως και με την πνευματική διάσταση που έχει η αίθουσά μας σήμερα ε, μπορούμε να ελπίζουμε πράγματι σε ένα θαύμα. Αλλά πάντως είναι τεράστια η πρόκληση και η δυσκολία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο, πρέπει να εξηγήσουμε ότι ουσιαστικά για του ανθρώπου του ίδιου μιλάμε. Αυτό μα απασχολεί. Σα ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την ομιλία. Θα ήθελα να ακούσω αν έχετε κάποια σχόλια, παρατηρήσει, ερωτήσει. Κάποιος από τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας ε, καλέσω επωνύμως να τοποθετηθείτε. Κύριε Σορβένη, κύριο Ζανάτο, θέλετε το λόγο. Κύριε Πυρίνσκι, ξέρω ότι εσείς θα αναλάβετε τα ενία περαιτέρω. Ε, θέλει όμως κάποιος από εσά να λάβει το λόγο. Κυρία Μαγκίνεση, νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς στην αρχή της συνεδρίας. Θέλουμε να συλλέξουμε περισσότερες ε, εντυπώσεις. Ναι, ευχαριστώ και ευχαριστώ που είστε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται και η φωνή των Ευρωβουλευτών. Αν όχι. Και οπωσδήποτε τα λόγια σας αντιχούν και θα τα ακούσουμε και πάλι ε, από τους επόμενους ομιλητές. Ίσως λοιπόν έχει νόημα να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Ο κύριος Σάβων ξέρω ότι θα έρθει σε λίγο, αλλά αναλαμβάνω εγώ να καθοδηγήσω το υπόλοιπο κομμάτι της συζήτησης. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια στο χώρο εργασίας, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το επόμενο θέμα. Συγκεκριμένη πτυχή θα συζητήσουμε σήμερα. Και μετά όσο είπε ο Λούκα για το ότι πολλοί είναι οι εργαζομένοι που δεν χαίρουν ανθρώπινης αξιοπρέπεια στο χώρο εργασίας, νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη επιλογή. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω την κυρία Σάνον Φόμαν και στο συγγνώμη για την προφορά από την Κάριτας της Ευρώπης υπεύθυνη πολιτικής και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης ε, αν θέλετε να αναλάβετε εσείς την καθοδήγηση των εργασιών και σε παρακαλώ Σάνον να ε, μιλήσετε για το θέμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στη δουλειά από την έποψη του εργαζομένου του ίδιου. Κυρία Φόμαν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σήμερα να μιλήσω ενώπιον σας εκ μέρους της Κάριτας της Ευρώπης με τους χαιρετισμού του Προέδρου που σκόπευε να έρθει να μιλήσει για λόγους όμως υγείας δεν μπόρεσε να έρθει στις Βρυξέλλες, να έρθει εδώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η Κάριτας της Ευρώπης είναι μία από τις επτά περιφέρειες της διεθνούς Κάριτας. Στην Ευρώπη 49 μέλη σε 46 κράτη έχουμε, άρα ξεπερνούμε το επίπεδο του Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ομάδα Επίση, προσπαθούμε να ενημερώνουμε πάντα και το Συμβούλιο της Ευρώπης για θέματα κοινωνικής πολιτικής, για την μετανάστευση, το άσυλο, ανθρωπιστική βοήθεια, κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Να ευαισθητοποιούμε πάντα. Έχουμε πάντως μια ενδιαφέρουσα προοπτική ούτως ε, που μας επιτρέπει να σχολιάσουμε την κατάσταση σχέση με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στην αγορά εργασίας και το ρόλο του κοινωνικού πυλώνα. Ωστόσο, πριν συνεχίσω θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό να επισημάνω ότι εκπροσωπούμε ή αναφερόμαστε στο άρθρο 11.2 και όχι στο άρθρο 17. Ε, δυνάμει αυτού βρισκόμαστε εδώ ε, και αυτό μας δίνει φωνή παρότι έχουμε συνεργασία με τις ε, εκκλησίες και παρότι η ε, διδασκαλία η θρησκευτική της Καθολικής Εκκλησίας είναι η πηγή έμπνευσής μας και ο οδηγός της εργασίας μας. Ας ξεκινήσω λοιπόν επισημένοντας ότι κάθε χρόνο κάνουμε έρευνες και μελέτες για την κατάσταση της φτώχειας, ιδιαίτερα των νέων φέτος, σε αυτούς αφιερώσαμε τη φετινή μελέτη. Και μάλιστα κοιτάξαμε λίγο πριν από την ε, ε, οικονομική κρίση του 2008, που διαπιστώσαμε ότι και πριν το 2008 ήταν δεκάδες εκατομμύρια οι νέοι που ζούσαν ε, κάτω από το επίπεδο της φτώχειας. Μετά την κρίση έχουν αυξηθεί τα ποσοστά, πολύ ψηλά τα νούμερα και το δυναμικό της φτώχειας, ο κίνδυνος να βρεθεί κανείς κάτω από το κατόφλι της φτώχειας. Διαπιστώνουμε ότι οι νέοι μετά την κρίση είναι πολύ πιο ευάλωτοι στη φτώχεια. Οι νέοι Ρωμά, οι νέοι με αναπηρίες, ε, ε, γυναίκες που μόνες τους αναθρέφουν τα παιδιά τους, ιδιαίτερα αν δεν έχουν πτυχίο, ε, γυναίκες και άνδρες από 16 έως 29 ετών με μεγάλες δυσκολίες στη μετάβαση από την ε, παιδική στην ε, ενήλικη ε, περίοδο της ζωής τους, δεδομένου ότι αυτούς έχει χτυπήσει περισσότερο και η ανεργία και οι συνθήκες εργασίας, τα συμβόλαια, οι συνθήκες απασχόλησης, η κοινωνική πρόνοια και οι συνθήκες αυτές. Ξέρουμε ότι πολλοί είναι οι νέοι που είναι παγιδευμένοι σε μακροχρόνια ανεργία, αλλά όχι μόνο νέοι. Χαρακτηριστικό και κύρια πηγή ανησυχία είναι η κακή ποιότητα και κακοπληρωμένε θέσει εργασία που άρα μπορεί κανεί να εργάζεται αλλά δεν μπορεί να κερδίσει αρκετά για να φτιάξει ένα μέλλον, για να φτιάξει οικογένεια. Ε, η μορφή της μαθητείας των ασκουμένων εξακολουθεί να επιτρέπει σε ένα νέο να ταξιδέψει από τη μία χώρα στην άλλη και να γνωρίσει κάτι καινούριο, αλλά χωρίς αμοιβή ή με πολύ ισχνή αμοιβή. Άλλα ζητήματα αφορούν τους μετανάστες υψηλής κατάρτισης και προσόντων που έχουν έρθει στην Ευρώπη, που, των, οποίων όμως αυτά τα προσόντα δεν αναγνωρίζονται, τουλάχιστον δεν αναγνωρίζονται στο, σε ισότιμο επίπεδο στην Ευρώπη και άρα χάνεται αυτή, η, αυτός ο πλούτος. Μεταναστευτικές κινήσεις διαπιστώνουμε και σε επίπεδο νέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή δεν υπάρχουν θέσει εργασία, Πολλοί είναι οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί νέοι που έχουν πάει στη Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρώπης, Ελπίζοντα ότι θα μπορέσουν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Η έκταση των συνεπειών της κρίσης ε, για τους νέους μπορεί να διαφέρει από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και οι νέοι τους έχουν τις πιο δυσμενείς συνθήκες να αντιμετωπίσουν και έτσι είναι πολύ πιο δύσκολο να εξασφαλίσουν ακόμη και την άσκηση κάποιων δικαιωμάτων τους. Είναι έντονες οι πιέσει, όλο και πιο έντονες την τελευταία δεκαετία που υφίστανται οι νέοι αυτοί και έχουμε να κάνουμε μια γενναία για πρώτη φορά που κινδυνεύει να ζήσει ζωή χειρότερη από ό,τι έχουν ζήσει οι γονείς της. Το μέλλον λοιπόν, το μέλλον και η αγορά εργασία, πώς μπορούμε αυτό να το εξασφαλίσουμε και ιδιαίτερα μέσα στι προοπτικές για το μέλλον της Ευρώπης και τις αλλαγές στην αγορά εργασία με την ψηφιοποίηση, με τα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια. με την ε, προσδοκία διαθεσιμότητας του καθενός ε, σε 24 ώρες βάση, ακόμα και αν το ωράριο εργασία του είναι από τι 9 τι 5 το βράδυ, θεωρούμε ότι μπορούμε να στείλουμε ανα πάσα στιγμή ένα email ή να πάρουμε ένα τηλέφωνο και να βρούμε ανταπόκριση αμέσω γιατί δουλεύει συνέχεια ο εργαζόμενο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά ζητήματα ανησυχητικά για του νέου, για το μέλλον, για την αγορά εργασία. Και κάτι το οποίο έχει ήδη απασχολήσει την κάρτα ε, της Ευρώπης από το 2016 είναι ο εντοπισμός βασικών αρχών για τη λειτουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος με βάση και τα κύρια χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού κοινωνικού συστήματος. Πυλώνες λοιπόν, τρεις πυλώνες η οικογένεια, θεμελιώδης πυλώνας ε, και στυλοβάτης της κοινωνίας και ως δίκτυα ασφαλείας, όπως έλεγα σε μια προηγούμενη συνάντηση που είχα σήμερα, όταν μιλούμε για κρίση απασχόληση, ξέρουμε ότι ο κόσμο θα γυρίσει πρώτα στην οικογένειά του και γενικά την κοινότητα μέσα στην οποία ζει για να εξασφαλίσει την υποστήριξη και αυτό κάπω προστατεύει από την ε, φτώχεια σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια τη χρηματοπιστωτική κρίση. οι ηλικιωμένοι σταξιούχοι ήταν οι μόνοι οι οποίοι είχαν ασφαλές εισόδημα και φρόντιζαν τους, ολόκληρη την οικογένειά του μέσα σε μικρά μάλιστα διαμερίσματα. Ο δεύτερο πυλώνα που σχετίζεται με τις αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβή είναι η αναγνώριση της συμβολής της ε, εργασίας στην κοινωνία και τις αξίες της. Εδώ λοιπόν ε, βοηθά η απασχόληση και στο να βρούμε το ρόλο μας και να δούμε την αναγνώριση του ρόλου μας ως ανθρώπων μέσα στην κοινωνία, ως προσώπων μέσα στην κοινωνία, να αναγνωριστεί ότι συμβάλλουμε και δουλεύουμε όχι μόνο για την οικογένειά μας αλλά για ολόκληρη την κοινωνία αυτή η συμμετοχή, η δημιουργία, η μέρημνα για τον εξωκόσμο κόσμο. Σημαίνει και συμμετοχή στην κοινωνία. Ο τρίτος πυλώνας, κοινωνική προστασία ως υγιής κοινωνική επένδυση. Οι τρεις πυλώνες λοιπόν περιλαμβάνουν το κοινωνικό μοντέλο της Κάριτας, ε, είναι μεταξύ τους σε σχέση αλληλεξάρτησης και συνεργασίας και βέβαια είναι ευθυγραμμισμένη με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα όπου περιγράφονται οι 28 αρχές και πρέπει να βρεθεί η σχέση, η συνάφεια μεταξύ τους γιατί το να εντοπιστεί μία αρχή και να λησμονηθούν οι άλλες δεν μπορεί να είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα ή παραγωγικό. Κοινωνικός πυλώνας λοιπόν Έχουμε μια σειρά από δραστηριότητε ευαισθητοποιήσει. Ήδη μιλήσατε για την προσπάθεια που έχουμε αναπτύξει για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική χρηματοδότηση για τον κοινωνικό πυλώνα. Γιατί παρά τι καλέ προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη δουλειά τη, ε, όταν πρότεινε ε, λύσει, ε, τελικά η πραγματικότητα μα φέρει αντιμέτωπου με τι επιλογέ των κρατών μελών όταν έρχεται η ώρα τη υλοποίηση των προτάσεων. Και βέβαια ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν ε, δύσκολες οικονομικές αποφάσεις, πρώτος που εξαφανίζεται είναι ο κοινωνικός πυλώνας. Κοινωνικές υπηρεσίες λοιπόν και έχουμε ετοιμάσει ε, έγγραφα που σας έχω φέρει κιόλα με προτάσεις για, τις τον κοινωνικό πυλώνα στην Ευρώπη, για, την, ε, για το συγκερασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου που μας έχει προσφέρει η Κάριτα της Γερμανίας και για θέματα ε, που ενδιαφέρουν πιστεύω τις θρησκευτικέ κοινότητες και ε, εκκλησίες. Στο μέλλον της Ευρώπης ε, έχουμε στις 27 Νοεμβρίου μία εκδήλωση από τις 9 έως τις 4 και 4, μία εκδήλωση της ΚΟΜΕΣΕ που θα ασχοληθεί ακριβώς με αυτές τις αλλαγές και το μέλλον της αγοράς εργασίας. Είμαι βέβαια ότι θα έχω και άλλο χρόνο για να απαντήσω σε ερωτήσεις και σταματώ εδώ για να καλωσορίσω και τον πρόεδρο επί τη ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η παρουσίαση του έργου της Κάριτας. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Και χαίρομαι που θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε όλα αυτά. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγική. Κύριε Σαμπόν, ε, ήρθατε την κατελότερη στιγμή. Εγώ δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων, οπότε είστε πολύ πιο κατάλληλος από εμένα για να συντονίσετε αυτή την ε, συζήτηση για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στον χώρο εργασίας. Έχουμε άλλους δύο ομιλητές που θα ακούσουμε. Έχετε τον λόγο πλέον να αναλάβετε το συντονισμό αυτής της συζήτησης, κύριε Σαμπον. Δυστυχώς πρέπει να φύγει και ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ. Σας ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Of Ήμουν και εγώ στην ΕΟΚΕ το, από το 1986. Κάθε φορά που τον συναντώ όμως ε, με εγκαταλείπει. Και συγχαρητήρια κύριε Πρόεδρε. Well, uh, I've been told I can speak in French. Μπορώ να μιλήσω γαλλικά από ό,τι ενημερώθηκα. Διάλογος των πολιτισμών λοιπόν και για χάρη του θα μιλήσω γαλλικά, έστω και αν η μητρική μου γλώσσα είναι η ισπανική. Αισθανόμαι καταρχάς βαθύτερη τιμή για την ε, πρόσκληση που μου ε, απευθύνθηκε και την ευκαιρία να ακούσω εσάς, να μοιραστώ μέσα σε αυτά τα λεπτά τα οποία εξέρουν και τιμούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον υψηλό αυτό οίκο. Μιλούμε για υψηλά ιδεώδη και αξίες ουσιοδέστατες. Και έτσι σε εμά τους πολιτικούς μερικές φορές υπενθυμίζεται και ότι είμαστε μεν παλιέ ε, παλιές καραβάνες όπως θα, λέγατε, θα λέγαμε, αλλά είμαστε ταυτόχρονα και ε, υπεύθυνοι και μέλη της κοινωνίας. Θα συντονίσω μόνο τη συζήτηση γιατί δεν θέλω εγώ να μιλήσω, αλλά να ακούσω. Συντονίσουμε λοιπόν το κομμάτι που αφορά την ε, αξιοπρέπεια στο, στην εργασία και μάλιστα στο χώρο εργασίας οι δύο διακεκριμένοι ε, σεβασμιότατοι ε, που έχουμε προσκαλέσει πιστεύω θα τοποθετηθούν και θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να το αναφέρω, ε, να τοποθετηθούμε όλοι, να είστε και εσείς συγκεκριμένοι στις, στους όρους εργασίας των εργαζομένων. Βέβαια όλοι δουλεύουμε έτσι, όλοι θα πούμε εργαζόμαστε, αλλά πώς το κρίνουμε το έργο το κρίνουμε όπως θα έλεγε μία μοναχή στο μοναστήρι που ενδεχομένως κάποιος απ' έξω να πει «Α, μια χαρά περνάει και είναι κλεισμένη μέσα στο μοναστήρι». Όχι, όλοι εργαζόμαστε, μιλούμε για, το, για τη δουλειά μας, μιλούμε για την εργασία, για το νέο που ετοιμάζεται να μπει στο χώρο εργασίας ε, μιας εργασίας πολλές φορές και εξαρτημένης ή εξαρτημένης από τα όσα έχει κάνει πιο πριν στη ζωή του. Θα μιλήσετε λοιπόν για τον εργαζόμενο και την αξιοπρέπεια του μισθωτού, του εργαζομένου σε εξαρτημένη εργασία. Εκείνο που έχει μια σχέση εξάρτησης, για να είμαστε απολύτω σαφείς. Άρα όχι για τη μοναχή μέσα, στον, ε, μέσα στο μοναστήρι. Όχι για μένα τη δουλειά που κάνω τώρα τουλάχιστον ως βουλευτής ή στο έργο που προσφέρουν οι ιερωμένοι, αλλά σε μια σχέση εξάρτησης μισθωτής εργασίας. Και εδώ μου έρχονται τα λόγια του Λακορντέρ και εκείνου μεγάλου θρησκευτικού, θρησκευτικής προσωπικότητας που έλεγε ότι ανάμεσα στον ισχυρό και στον αδύναμο η ελευθερία διακρίνει ο νόμος εξισώνει, φέρνει σε ίσους όρους. Και αυτό είναι απολύτως αληθές. Απολύτως αληθές γιατί μιλούμε τελικά για αξιοπρέπεια. Μιλούμε για κυριαρχή θέση, φαντάζομαι θα αναφερθείτε και εσείς. Μιλούμε για αξιοπρεπή μεταχείριση, για σεβασμό στην αξιοπρέπεια. Και γιατί. γιατί στην Ευρώπη, και πιστεύω με κάποιες ίσως εξαιρέσεις μόνο, αλλά πάντως ο νόμος έχει φέρει αποτελέσματα απτά και αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι βεβαίως να προσαρμόσουμε τον νόμο στις σύγχρονες συνθήκες εργασίας, στον εξυγχρονισμό, την τεχνολογία. Αλλά ο νόμος έχει φέρει αυτή την ελάχιστη έσως, αυτό μίνιμουμ της αξιοπρέπειας. Βεβαίως όλα μπορούν να βελτιωθούν. Άρα από τι εξαρτάται μερικές φορές η αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου στο χώρο εργασίας του. Δεν νομίζω ότι όσοι έχει, είσαστε εδώ σήμερα θέλετε να αναφερθείτε στην αξιοπρέπεια που προσφέρει ένας ε, ικανοποιητικός μισθός, που βεβαίως είναι πολύ σημαντικός, αλλά που θα συζητηθεί σε ένα άλλο πάνελ. Εμείς μιλούμε για αξιοπρέπεια σε όρους εργασίας, σε αξιοπρέπεια μετά και μέσα στην ε, πραγματική ζωή, όπως είπαμε, δηλαδή να μην είναι κανείς φτωχός, αλλά εδώ μιλούμε για την αξιοπρέπεια στον χώρο εργασίας. Από τη στιγμή λοιπόν που αρχίζουν οι νόμοι να φέρουν τα αποτελέσματά τους και που αρχίζουν να προσαρμόζονται στην ε, καινοτομία, στην εξέλιξη, την τεχνολογική, πρέπει να κοιτάξουμε πώς αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος και, και τα προσωπικά του στοιχεία Πολλές φορές εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν μισθωτό που μπορεί να είναι επικεφαλής μιας ομάδας και έναν άλλο μισθωτό που όμως είναι απλώς μέλος της ομάδας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την σχέση αυτήν και των, των δύο αυτών μισθωτών μεταξύ τους που όμως είναι σχέση ιεραρχίας και σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί η αξιοπρέπεια που θα κρίνουμε εδώ έτσι λοιπόν στους τους ε, προσκεκλημένους μας θέτω το εξής ερώτημα, όπως και σε εσά άλλωστε, να κοιτάξουμε τη ρίζα της αξιοπρέπειας του χώρο εργασίας. Μήπως είναι μια αξιοπρέπεια η οποία εν τέλει θα εξαρτηθεί από αντιλήψεις, αξίες, παιδεία. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι οι πνευματικές αξίες, οι θρησκείες δηλαδή, είναι σεβασμό ότι οι προσκεκλημένοι δεν ανήκουν στη δική μου θρησκεία, ούτε και θα μπορούσαν να ανήκουν γιατί εγώ δεν έχω θρησκεία. Αλλά και ο αγνωστικιστής γνωρίζει την ηθική. Έτσι λοιπόν, στο σημερινό κόσμο, όταν έχουμε να κάνουμε με νόμους που ξέρουμε ότι δεν είναι ποτέ επαρκείς, επιμένω και το υπογραμμίζω, όταν εξετάζουμε όμως ένα νόμο έστω επαρκή ή τον εξετάζουμε ως επαρκή, δεν πρέπει να αναφερόμαστε σε αξίες όπως η παιδεία που ανέφερα νωρίτερα. Και χωρίς να θέλω να σας καθυστερήσω περισσότερο, ήθελα να θέσω αυτό το ερώτημα προς ανάπτυξη. Γιατί έχουμε αξίες που κανένας νόμος του κόσμου δεν θα μπορέσει να κωδικοποιήσει στην πράξη. Μετά, τα πάντα θα εξαρτηθούν από το πρόσωπο. Ζητώ συγγνώμη που χρειάστηκα αυτά τα 5-10 λεπτά για αυτή την ε, ε, εναρκτήρια εισήγηση. Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω πρώτα τον μουφτή, τον σεβασμιότατο ε, Ιγνάτιο, τον σεβασμιότατο. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης λοιπόν από την Ορθόδοξη πίστη και ζητώ συγγνώμη για την ε, ε, προφορά τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο. Καλό, εμείς το Ιγνάτιο, το έχουμε σαν όνομα στην Ισπανία, ο Ιγνάτιο Λογιόλα άλλωστε είναι πολύ γνωστός. Ε, ο Μητροπολίτης λοιπόν Ιγνάτιος, Μητροπολίτης Δημητριάδος και Ελμυρού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Γεννηθεί το 56 στην Αθήνα, νεότερος από μένα, δεν σας πω πόσο όμως ο νεότερος, μέλος πολλών ε, επιτροπών της Συνόδου, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκπροσωπεί την ε, ε, Εκκλησία της Ελλάδος στο Μεγάλο Συμβούλιο των Ορθοδόξων Εκκλησιών που έλαβε χώρα στην Κρήτη πριν από δύο χρόνια και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Board of Directors της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών του Βόλου. Ταυτόχρονα είναι πολύ γνωστός και στα Ερτζιανά. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω και στα δίκτυα, τα διαδίκτυα. Είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει στην κοινωνία. Πιστεύει στη διαρκή επικοινωνία. Και παρουσίασε από το 1992 το 2013 ένα ε, πρόγραμμα στην ελληνική τηλεόραση με πολύ μεγάλη επίχυση και, θέμα, απήχηση και θεαματικότητα, ε, με πολλές ε, ομιλίες και παρουσίασεις για θέματα της καθημερινής ζωής και της πνευματικής μαζί. Καλύτερο εκπρόσωπο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που άλλωστε βρίσκεται στην ουσία της θρησκευτική του πίστης δεν θα μπορούσαμε να έχουμε προσκεκλημένο εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, σεβασμιότατε που είστε εδώ. Περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία την δική σας παρέμβαση και θα σας παρακαλούσα ή δυνατόν να <laughs> περιοριστείτε στα 8 λεπτά. Εάν περιοριστείτε δεν θα είναι αμαρτία, εάν τα τηρήσετε δεν θα θυμώσω. Thank you very much, Mr. President. I will speak Greek, so you need translation. Thank you. Η περάσπιση της αξιοπρέπειας των τέκνων του Θεού στη ζωή και την εργασία – Ξεκινώντα την τοποθέτησή μου, θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώ και τον Γενικό Γραμματέα τη Συνόδου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, για την τιμητική αυτή πρόσκληση που μου δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σα και να μοιραστώ σκέψει και προβληματισμού για ένα όντω φλέγον θέμα, όπω αυτό του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και του ρόλου των θρησκευτικών παραγόντων στην εφαρμογή του. Θα ήθελα βέβαια εξ αρχή να διευκρινίσω ότι δεν είμαι ειδικό των ευρωπαϊκών θεμάτων ούτε των εργασιακών σχέσεων. Είμαι ένα απλό χριστιανό Ορθόδοξο Επίσκοπο, δεσμευμένο στο ευρωπαϊκό όραμα, ο οποίο προέρχεται από μια χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου, την Ελλάδα. Μια χώρα η οποία βρέθηκε πολλέ φορέ για αρνητικού δυστυχώ λόγου τελευταία στο επίκεντρο τη επικαιρότητα. Γι' αυτό και θα μιλήσω για το νευραλγική σημασία υποσυζήτηση θέμα ω απλό επίσκοπο και επιμένα και όχι ω τεχνοκράτη ή ειδικό των ζητημάτων. Αυτό είναι νομίζω τελικά και το ζητούμενο από εμένα. Τι έχει να πει από τη δική του σκοπιά ένα θρησκευτικό λειτουργό, με την ευθύνη μια θρησκευτική κοινότητα, ορθόδοξη χριστιανική εμπροκειμένου, για τι αξιοπρεπεί συνθήκε εργασία για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, αλλά και ευρύτερα για την κοινωνική συνοχή και το μέλλον τη κοινωνική Ευρώπη. Επιτρέψτε μου στο ξεκίνημα τη τοποθέτησή μου να θυμίσω ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε ταπεινά και έζησε ταπεινά, Συναναστρεφόμενο συχνά ανθρώπου των κατώτερων κοινωνικά τάξεων, ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Ο ίδιος, αν και ιό του Θεού, άσκησε από μικρό το χειρονακτικό επάγγελμα του μαραγκού, ενώ πολλοί από του μαθητέ του ήταν απλοί ψαράδε και μάλιστα του γλυκού νερού. Είναι επίση χαρακτηριστικό ότι στου λόγου και τι παραβολέ του συχνά αναφέρεται σε βοσκού και επιμένε με του οποίου παρομοιάζει τον εαυτό του και την αποστολή του. Ενώ σύμφωνα με τι ευαγγελικέ διηγήσει για τη γέννησή του, βοσκοί την αναγγέλουν και τη δοξολογούν. Με άλλα λόγια, ευθύ εξ αρχή, οι ευαγγελικέ μαρτυρίε για τον Ιησού Χριστό εισάγουν την ιερότητα αλλά και την αξιοπρέπεια τη εργασία, όσο ταπεινή και αν είναι αυτή. Μια ιερότητα και αξιοπρέπεια που πηγάζουν από την μοναδικότητα τη θεμελιώδη ερώτητα και αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπινου προσώπου που σύμφωνα με τη χριστιανική αντίληψη είναι εικόνα του ζώντος Θεού. Γι' αυτό και κάθε ανθρώπινη εργασία και έργο και όχι μόνο τα λεγόμενα πνευματικά σε εισαγωγικά έχουν σημασία για την καταξίωση και σωτηρία του ανθρώπου και όλου του κόσμου. Αναλαμβάνοντας με την ενσάρκωση του ο Υιός και Λόγος του Θεού όλη την ανθρώπινη φύση και ιστορία, κάθε πλευρά και κάθε πτυχή της ζωής μας αναλαμβάνει και μεταμορφώνει και τον ανθρώπινο μόχθο, την εργασία και το επάγγελμα, υπερβαίνοντας εκείνη την αντίληψη που τα θέλει να είναι μέσα μόνο πλουτισμού και ικανοποίηση ατομικών, εγωιστικών αναγκών και επιθυμιών και μεταποιώντας τα με την έμπρακτη αγάπη και αλληλεγγύη σε αφορμή και μέσα κοινωνίας με τον συνάνθρωπο και το Θεό. Γι' αυτό και στη χριστιανική αντίληψη δεν έχουν θέσει στάσεις και κατανοήσεις που αμαυρώνουν έστω και στο ελάχιστο την εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Αντιλήψεις και συμπεριφορές που εργαλειοποιούν το ανθρώπινο πρόσωπο και το υποτάσσουν σε αλότρια συμφέροντα, λησμονώντα ότι ούτε πάρτο μόνο ζήσει άνθρωπος. Και ότι όπως το Σάββατο, έτσι και η εργασία ή η οικονομία έγιναν για τον άνθρωπο και όχι το αντίστροφο που δυστυχώς συμβαίνει πολλές φορές στην εποχή μας. Είναι χαρακτηριστικό σε σχέση με τα παραπάνω οι συμπεριφορέ απαξίωση και εκμετάλλευση εργασία του πλησίων και μεροληψία σε βάρο των φτωχών αποδοκιμάζονται ρητό στη χριστιανική παράδοση. Η επιστολή Ιακώβου στην Καινή Διαθήκη μιλάει με σκληρά λόγια για την αποστέρηση του μισθού των εργατών. Ενώ μεταγενέστεροι διδάσκαλοι και πατέρε τη Χριστιανική Εκκλησία καταδικάζουν με αυστηρότητα ανάλογε συμπεριφορέ όπω και διακρίσει με βάση το φύλλο ή τη φυλή την κοινωνική, την πολιτισμική προέλευση κλπ. Στα κείμενα πολλών πατέρων της Εκκλησίας προβάλλεται μάλιστα η ιδέα της ιερότητας των πτωχών, που θεωρούνται οι κατεξοχήν φίλοι του Θεού. Έτσι η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη το συμπάσχην και συνοδύνει με τα θύματα της ιστορίας δεν αποτελεί για το χριστιανό ένα καθήκον απλώς μεταξύ πολλών άλλων, το οποίο υποχρεούται να εκπληρώσει προκειμένου να επιτύχει την έννοια του Θεού κατά την ημέρα της μέλουσας κρίσης, αλλά συνιστά τον τρόπο ζωής που μας έδειξε ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ρητός μας δίδαξε να αναγνωρίζουμε το πρόσωπό Του στο πρόσωπο των ελαχίστων αδελφών μας, στο πρόσωπο του κάθε πλησίον, του φτωχού, του πεινασμένου, του ξένου, του περιθωριακού, του μετανάστη. Δεν χρειάζεται στην προκειμένη περίπτωση παρά να φέρουμε στο νου μας τα πολύ γνωστά βιβλικά παραδείγματα του καλού Σαμαρίτη και της μέλουσας κρίσης για να αποκτήσουμε μια επαρκή εικόνα του πώς εννοείται στη χριστιανική προοπτική η αγάπη, η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη. Όπως έγραφε ο Ρώσος χριστιανός φιλόσοφος και επαναστάτης Νικολάη Μπερδιάγεφ, απηχώντας εν προκειμένου το πνεύμα αλλά και το γράμμα των καθολικών επιστολών του Ιακώβου και του Ιωάννη. Το να παλεύω για το ψωμί μου είναι πρόβλημα υλικό, αλλά το να παλεύω για το ψωμί του διπλανού μου είναι πρόβλημα πνευματικό. Οι μεγάλοι πατέρε τη Εκκλησία καταδίκασαν απερίφραστα επίση την εκμετάλλευση τη εργασία και τη συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των ολίγων, καθώ και την κοινωνική αδικία την οποία αρνήθηκαν να αποδεχτούν ω θέλημα του Θεού. Προερχόμενο λοιπόν από μια τέτοια θρησκευτική και πνευματική παράδοση, δεν μπορώ παρά να χαιρετήσω με ικανοποίηση και να θεωρήσω πολύ σημαντικά βήματα προ τη σωστή κατεύθυνση τα όσα ο Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων προβλέπει για το θέμα που μα απασχολεί. Και μάλιστα τα σχετικά με τι αξιοπρεπεί και ασφαλεί συνθήκε εργασία, την κοινωνική προστασία και την προστασία τη υγεία και τη ασφάλεια στην εργασία, το επίπεδο αμοιβών και αξιοπρεπού διαβίωση, την αποτροπή τη φτώχεια των εργαζομένων, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και προσωπική ζωή και άλλα. Χωρί να θέλω επουδενή να ακυρώσω την πρόοδο που αντιπροσωπεύουν οι παραπάνω προβλέψει, δεν θα μπορούσα να μην επισημάνω και εγώ αυτά που ήδη ελέγχθησαν, ότι αυτές πόρο απέχουν από την πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα πολλοί λαοί στην Ευρώπη, όπου η ελαστικοποίηση και η προσωρινότητα των μορφών εργασίας, η κατάχρηση των άτυπων συμβάσεων και η φτωχοποίηση ολοένα και μεγαλύτερων στρωμάτων του πληθυσμού κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Αν δεν στραφώ στην περίπτωση της χώρας μου, της Ελλάδος, που δοκιμάζεται τα τελευταία 8 χρόνια από τη βαθιά οικονομική κρίση τη μαζική ανεργία ιδιαίτερα των νέων, τα όλο και μεγαλύτερα κύματα μετανάστευση στο εξωτερικό και τη διαρροή εγκεφάλων μορφωμένων, την έξαρση του μεταναστευτικού και προσφυγικού προβλήματο, την κατάρρευση του συστήματο υγεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε μεγάλο βαθμό, την αχρήστευση των συλλογικών συμβάσεων σε πολλέ περιπτώσει και την εντυνόμενη ελαστικοποίηση των μορφών εργασία, του μισθού πείνα και τη φτωχοποίηση τη άλλοτε ευημερούσα μεσαία τάξη, επίση τη δημογραφική κρίση, την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των αστέγων και εν γέννη όλα όσα θυμίζουν αυτό που θα ονομάζαμε ανθρωπιστική κρίση, τότε οι κατά τα άλλα θετικές προβλέψεις και πρόοδοι του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων μοιάζουν δυστυχώς με κενό γράμμα και ευχολόγια που δεν φαίνεται να απαντούν στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών της Ευρώπης και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, καθώς βρίσκονται σε πλήρη αναδυστυχία με την ολοένα επιδεινούμενη πραγματικότητα που οι πολίτε τη Ευρώπη βιώνουν σήμερα. Για την υπέρβαση τη αντίφαση μεταξύ ωραίων λόγων και θλιβερή πραγματικότητα, μεγάλη σπουδαιότητα αποδίδεται στα μέσα και τα μέτρα εφαρμογή των όσων προβλέπει ο Ευρωπαϊκό Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων, καθώ και στην εγγραφή στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, όπω ήδη ελέγχθη, σχετικών κονδυλίων για την εμπέδωση, υλοποίηση και εφαρμογή των προβλέψεων αυτών. Όπω τονίζεται και σε σχετικέ παρεμβάσει του Χριστιανικού Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ευρωδιακονία, το βασικό ερώτημα είναι πώς οι αρχές του κοινωνικού πυλώνα, οι οποίες δεν είναι εκτελεστές, μπορούν να μεταφραστούν σε σημαντικές κοινωνικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και πώς οι προβλέψεις και οι πρόνοιες του πυλώνα αυτού δεν θα μείνουν ανενεργές, όπως συνήθως συμβαίνει με άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες που απέβλεπαν στην οικοδόμηση μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης. Αγαπητοί μου, νομίζω πω πάνω απ' όλα αυτό που πρέπει να γίνει συνείδηση και στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων είναι το ότι διακυβεύεται σε σχέση με το μέλλον τη Ευρώπη. Το τι διακυβεύεται. διακυβεύεται. Εάν λοιπόν το ευρωπαϊκό όραμα θέλει να ανακτήσει τη δυναμική και την έγκλη του, καθώ και την ικανότητά του να συνενώνει και συνεγείρει ανθρώπου διαφορετικών καταβολών, τότε οφείλει να υπερβεί την κυρίαρχη σήμερα αντίληψη μια Ένωση που προσδιορίζεται από οικονομικού κανόνε και μέτρα λιτότητας. Όπω έχει ήδη επισημανθεί σε κείμενο του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών με τίτλο «Πέρα από την ευημερία», δεκαετίε πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγενίασε τη λειτουργία της ως ένα εμπνευσμένο έργο ειρήνης και καταλλαγής. Ενώ από την αρχή της λειτουργίας της η πρωταρχική κινητήρια δύναμη για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η επίτευξη στόχων με σαφώς ευρύτερο περιεχόμενο από αυτό της οικονομικής συνεργασίας. Αυτή η ρωμαλαία δήλωση επαναφέρει στο νου μα την ιστορική διακήρυξη των Ευρωπαϊκών Χριστιανικών Εκκλησιών το 2001, σύμφωνα με την οποία χωρί κοινέ αξίε η ενότητα δεν θα διαρκέσει. Ερχόμαστε έτσι αντιμέτωποι με το κρίσιμο ζήτημα των κοινών αξιών, καθώς και με το όραμα των θεμελιωτών ή των ξεχωριστών ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jack Delors, ο οποίο υποστήριξε ότι δεν θα πραγματώσουμε το όραμα για την Ευρώπη βασιζόμενη αποκλειστικά και μόνο στη νομική πραγματογνωμοσύνη ή την οικονομική επάρκεια. Εάν δεν καταφέρουμε να δώσουμε ψυχή στην Ευρώπη, τότε θα αποτύχουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Euh, Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο και δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό να σχολιάσω πόσο πολύ συμφωνώ με τα άγια λόγια του, έτσι θα το πω, πόσο προφανές είναι αντίθετα με αυτό που ορισμένοι σήμερα ισχυρίζονται, όπως κάποιος πρωθυπουργός που πρόσφατα επεσκέφθη το Στρασβούργο και είπε ε, καλά ευρωπαϊκή ε, κοινωνική Ευρώπη, σιγά δεν υπάρχει κιόλα ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Όχι, όχι, δεν αληθεύει αυτό. Από την εποχή των ιδρυτών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, διαφοροποιείται από, τους άλλους, από τις άλλες υπήρους και την Αμερικανική παραδείγματι, γιατί θεμελιώνεται πάνω και στην οικονομική συνεργασία και την ηθαγένεια, την κοινωνική Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι στι ιδρυτικέ συνθήκε ιδρύεται αυτό το οποίο δεν, έχουν, δεν γνωρίζουν οι ΗΠΑ, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που ο πρόεδρος καθόταν εδώ δίπλα μου μόλι τώρα. Και είπε, ε, είπαν οι ιδρυτέ λοιπόν από την πρώτη στιγμή, βεβαίω να γίνει οικονομική συνεργασία. Αλλά αν οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμφωνούν, δεν θα φέρει αποτέλεσμα από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό ιδρύθηκε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Και ευχαριστώ θερμά το Σεβασμιότατο Ιγνάσιο, ο οποίος ε, έθεσε έτσι με τα σοφά του λόγια, με την Αγία Σοφία του την ε, βάση αυτής της συζήτησης. Η Ευρώπη ή θα είναι κοινωνική ή δεν θα είναι Ευρώπη. Είμαι πεπισμένο γι' αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτά τα θερμά λόγια. Σεβασμιότατε. Και έχω τώρα την τιμή να παρακαλέσω τώρα τον κύριο Νέτζ Μιντάμποφ από τη Βουλγαρία, μέγα μουφτή της περιοχής της, του Σμόλιαν της Βουλγαρίας. Είναι ασφαλώς πολύ πολύ νεότερος από μένα ο κύριος Ντάμποφ, έχει αυτή την τύχη, δεν θα σας πω όμως την ηλικία του. Γεννήθηκε στην ίδια την ε, επαρχία του Σμόλια, στην ε, Βουλγαρία, του Σμολιάννα, εκεί ακριβώς όπου υπηρετεί, εκεί και πήγε σχολείο, εκεί σπούδασε στο Μάνταμ, Μαντάνα, Μάνταν ή Μάνταν στα γαλλικά. Ήταν ε, ιερωμένο, είπαμε, στο Μπόριε, στην περιοχή του πάλι, το χωρίς το οποίο γεννήθηκε, μετά ανέλαβε καθήκοντα ε, γερωμένου στο ίδιο το Σμόλιαν, συνεχίζοντας τις Ισλαμικές σπουδέ στο Ινστιτούτο της Σόφιας, από το οποίο αποφύτησε, ε, υπηρέτησε ως σύμβουλος για θρησκευτικά θέματα στο Δημαρχείο του Ριουντοζέμ. Και ανέλαβε καθήκοντα μέλους του, ΥΠΑ, ε, του Θρησκευτικού Συμβουλίου της Βουλγαρίας, εκπροσωπώντας το Σμόλιαν, την περιοχή του, όπου και σήμερα ακόμη υπηρετεί ως μουφτής. Έχει πολύ ευρύτερη από ό,τι έχω ε, θεώρηση της ε, κοινωνίας ε, και του ανθρώπου είναι παντρεμένος. Εγώ μπορώ να συγκριθώ μαζί του γιατί τον έχω ξεπεράσει τρεις φορές, αλλά επιπλέον έχει και παιδιά, δύο παιδιά που εγώ δεν έχω. Αυτή λοιπόν η ανθρώπινη διάσταση αλλά και η βαθιά του κουλτούρα, οι βαθιές του ουμανιστικές ανθρωπιστικές γνώσεις και η θρησκευτική του καλλιέργεια νομίζω θα του επιτρέψουν να μας μιλήσει για τις αξίες της θρησκείας και της αξιοπρέπειας στον χώρο εργασίας. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ θερμά την ε, κυρία Μάρια Μαγκίνες, πρώτη αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι εδώ σήμερα. Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των θρησκειών και δογμάτων, κυρίες και κύριοι, ο κοινωνικός πυλώνας, ο ρόλος των εκκλησιών ο ρόλος της θρησκευτική πίστης. Θα ήθελα να απευθύνω τους χαιρετισμού του Μέγα Μουφτή της Βουλγαρίας, τον οποίο εκπροσωπώ σήμερα, για να σας παρουσιάσω μία έκθεση για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στον χώρο εργασίας. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι κομμάτι της ανθρώπινης προσωπικότητας. Χωρίς αξιοπρέπεια δεν είναι άνθρωπος ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος υφίσταται διακρίσεις, απόρριψη, περιθωριοποίηση. Δεν είναι ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Το Ισλάμ θεωρεί ότι η αξιοπρέπεια είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρωπινής προσωπικότητας. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι παιδιά, είναι τέκνα του Θεού. Ο οποίος Θεός είπε «Άνθρωποι σας έφτιαξα από τον άνδρα και τη γυναίκα ανεξαρτήτως της φυλής, του φίλου, της κοινωνικής προέλευσης, της θρησκείας, της εθνικότητας, της ευαγένειας του κοινωνικού ε, καθεστώτος, της κοινωνικής τάξης, πρέπει ο άνθρωπος να χαίρει του σεβασμού των άλλων. Γιατί είναι το πλέον ιερό «ον» που δημιούργησε ο πλαστουργός. Και ο ένας άνθρωπος οφείλει να σέβεται τον άλλο, γιατί του σέβεται όλους ο Θεός. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια λοιπόν είναι αξία αναπαλωτρίωτη και αδιαπραγμάτευτη. Όπως άλλωστε καταγράφεται και στον ε, χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και στην Οικονομική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι η εργασία για το Ισλάμ μια ιερή πράξη. Χάρη σε αυτήν ο άνθρωπος εξασφαλίζει την αξιοπρέπειά του, ξεφεύγει από τη φτώχεια, δουλεύει, εργάζεται για την οικογένειά του, αλλά και το καλό της κοινωνίας του. Ο νομεθενισμός θέλει να εξασφαλίσει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Είτε είναι μισθωτός, είτε είναι στέλεχος, είτε είναι αφεντικό ή προϊστάμενος. Ο προϊστάμενος ή το αφεντικό θα πρέπει να προσφέρει δουλειά αντίστοιχη στι δεξιότητες του εργαζομένου. Και ο εργαζόμενος πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια, αλλά και να, εργάζεται, να έχει τη δυνατότητα να εργάζεται σε συνθήκες αγαστές στο χώρο εργασίας. πρέπει να την χάνει του σεβασμού της ε, ιεραρχίας των προϊσταμένων του με μια ευκαιρία και δυνατότητες για διαρκή επιμόρφωση. η ανθρώπινη πόρη. ως υπηρεσία πρέπει να αναπτύσσουν το δυναμικό των εργαζομένων. Πώς όμως ο προϊστάμενος, το στέλεχος θα ε, δώσει κίνητρα για ανάταση στον εργαζόμενο. Αυτό νομίζω επιτυγχάνεται κατά τον καλύτερο τρόπο με την αξία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όταν μιλούμε για ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μιλούμε για έναν άνθρωπο που ολοκληρώνεται σαν προσωπικότητα μέσα στην κοινωνία, που βρίσκει τη θέση του και τιμά την κοινωνία στην οποία ζει. Δεν πρέπει κανείς να υποχρεούται να κάνει επιλογή μεταξύ της κοινωνίας του, της συμμετοχής του στην κοινωνία και το γίγνεσθε και την, και την ε, δική του ανέλυξη. Εάν κανείς δηλαδή είναι περιθωριοποιημένος, δεν μπορεί να σταθεί μέσα στο χώρο εργασίας. Πρέπει να εξασφαλιστεί ένα περιβάλλον εργασίας ευχάριστο, ένα περιβάλλον με ηρεμία και ε, καλές συνθήκες για όλους τους εργαζομένους. Η δάλος και η ε, επιχείρηση θα έχει χάσει και η κοινωνία η ευρύτερη θα έχει χάσει όπως και ο εργαζόμενος. Έχουμε λοιπόν εδώ το κλειδί των ε, κινητήριο μοχλό της ε, επιχείρησης όπως και της κοινωνίας στο πρόσωπο του εργαζομένου. Και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί μια ισορροπία μεταξύ ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου μέσα στην Ευρώπη που, θα, που θέλει να είναι γνήσια κοινωνική. Κάθε ένας έχει δικαίωμα σε ελευθερία, σε αξιοπρέπεια, σε συνθήκες εργασίας που του επιτρέπουν να αναπτύσσει το δυναμικό του και τη δημιουργικότητά του την μέρα που θα μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε αυτό, μπορούμε να μιλούμε πλέον για ευημερία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ θερμά. Σα ευχαριστώ. Σε μας θίξατε μια πτυχή που περίμενα να ακούσω από εσά Από έναν από τους προσκεκλημένου μας. Αξιοπρέπεια στο χώρο εργασία, η οποία αλλά και γενικότερα η αξιοπρέπεια, η οποία στηρίζεται στον σεβασμό. Πράγμα όχι εύκολο βέβαια. Και είπατε ότι είναι δύο οι όψεις του νομίσματος και ότι πρέπει να πετύσουμε το σεβασμό του ανωτέρου προς τον υφιστάμενο αλλά και βέβαια του υφισταμένου το σεβασμό να απαιτήσουμε για την αξιοπρέπεια του προϊσταμένου. Ο σεβασμός λοιπόν και τώρα έρχεστε εσείς στο προσκήνιο για να μας επιτεθείτε και στους τρεις γιατί η κυρία ε, δίπλα μου έδειχνε κάπως να αποστασιοποιείτε όχι δεν ε, είσαστε στο απειρόβλητο μπορείτε να μας ε, απευθύνετε τραβέλη σας και εγώ ξέρετε ότι μπορώ να γίνω και πολύ προκλητικός και ε, κακός εντό εισαγωγικών. Θα ήθελα λοιπόν πάρα πολύ να μας πείτε, ξεκινώντας τις δικές σας ε, ε παρεμβάσεις, με κάποια ερώτηση που πάντα ξέρω ότι είναι πολύτιμη και εύστοχη. ποιο. θα ήθελε παρακαλώ να λάβει το λόγο, δίνοντας κιόλας... Ε, συστηνόμενος κιόλας δίνοντας τα στοιχεία του για να ξέρουμε ποιον εκπροσωπεί, ποιος θέλει να ξεκινήσει και όχι όλοι μαζί παρακαλώ. Παρακαλώ. Θα μπορούσα να μιλήσω ισπανικά. Θα σας καταλάβω εγώ, λέει ο κύριος Σαμπόν. οι υπόλοιποι θα δούμε. Ναι. Κάρλος ε, Σαρία από την Ισπανία, από τους ε, σοσιαλιστές χριστιανούς και μέλος των, της οργάνωσης των Διεθνών Σοσιαλιστών Χριστιανών. Είναι πολύ σημαντικό να συζητούμε την, το ρόλο του χριστιανισμού, των χριστιανικών οργανώσεων από την κοινωνική πλευρά, ε, όχι μόνο από την πλευρά των ελευθεριών, όπως είπε η Αντιπρόεδρος. Και νομίζω ότι αυτό το πάνελ είναι πολύ σημαντικό, γιατί Πολύ συχνά μιλούμε για τη συμβολή των θρησκειών από τη σκοπιά του πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, για παράδειγμα. Αλλά δεν ασχολούμαστε επαρκώς με το ρόλο των θρησκειών στην καρδιά της οικονομίας, των παραγωγικών σχέσεων, των επιχειρήσεων. Και επειδή μιλούμε εδώ για την αξιοπρέπεια στον χώρο εργασίας και την, τις αξιοπρεπείς αμοιβέ, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας το τι γίνεται στους χώρους εργασίας. Θέλω να υπενθυμίσω αυτό που είχε πει και ο Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος σχετικά με την αξιοπρέπεια στον χώρο εργασίας. και το προβάδισμα που πρέπει να έχει εργασία έναντι του κεφαλαίου. Αυτό βεβαίως δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής εδώ στη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο της συζήτηση που πρέπει να γίνει. Ο στόχος της ε, οικονομίας με την κυριαρχία του, του κεφαλαίου είναι αυτό που δημιουργεί πολλά από τα προβλήματα που έχουμε. Χρειαζόμαστε μια πιο παραγωγική οικονομία που θα θέτει στο επίκεντρό της τους ανθρώπους πολύ περισσότερο από ό,τι το κάνει σήμερα. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση και τη διεύθυνση των εργαζομένων αλλά και την ε, επίτευξη των αποτελεσμάτων που αποφέρουν αυτές οι επιχειρήσεις. Συμμετοχή τους δηλαδή στην ίδια τη διακυβέρνηση των ε, επιχειρήσεων μέσω διαφόρων μορφών, ε, αν θέλετε, κεφαλαίου. Εγώ προέρχομαι από τη χώρα των Βάσκων και εκεί υπάρχει μια πολυεθνική εταιρεία, η Μανδραγών, η οποία ιδρύθηκε από ιερέα ο οποίος εφάρμοσε τις το, το χριστιανικό δόγμα. Η επιχείρηση αυτή έχει περάσει από μια μεγάλη κρίση. Κατασκευάζει οικιακές συσκευές. Ωστόσο, παρά την κρίση, επέλεξε να μην απολύσει τους εργαζόμενους, ώστε να δώσει ε, κέρδη στους μετόχους της. Αντιθέτως, η Μοντραγόν ε, δημιούργησε ένα αποθεματικό 50 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε ακόμη και αν χρεοκοπούσε να ήταν εξασφαλισμένη η εργαζόμενή της. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό και θετικό παράδειγμα για το πώς πρέπει να γίνεται η διοίκηση μιας επιχείρησης. Και τέλος αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που υπόθηκε και νωρίτερα, αυτή η διαδικασία της ε, ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης, όλα αυτά προκαλούν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στους χώρους εργασίας, γιατί υπάρχει όλο και μεγαλύτερη παραγωγικότητα χωρίς έμπρακτη ανθρώπινη παρέμβαση. Αν θέλουμε λοιπόν τα μοντέλα της οικονομίας να είναι βιώσιμα, πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό πώς η βελτίωση της και η αύξηση της παραγωγικότητας στην πραγματικότητα θα πρέπει να απελευθερώνει τον ε, ελεύθερο χρόνο, να διευρύνει τον ελεύθερο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους οι άνθρωποι, αλλά όχι εις βάρος τους μέσω των εργασιακών σχέσεων που θα τους επιβληθούν. Και αυτό είναι κάτι που αφορά όλους τους, ε, ό, όλες τις ομολογίες, όλες τις θρησκείες. Ε, μου ε, επαναλαμβάνετε παρακαλώ την ερώτηση. Α, δεν ήταν ερώτηση. Λοιπόν, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λέει ο πρόεδρος για ε, για όλη την παρέμβαση. Γνωρίζω αρκετά καλά τη Μοντραγκόν, αυτή την συνεταιριστική οργάνωση στην οποία αναφερθήκατε. Συστήθηκε από αυτόν τον οποίο θεωρώ δάσκαλό μου στην πολιτική και το συνδικαλισμό. Ναι, ναι, μεταφράζεστε, μεταφράζεστε, κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα να ακούσουμε και άλλους, παρακαλώ, από τους παρευρισκομένους. Και στο θέμα της ε, σπατάλης ε, που ανέφερε και ο Παπας Φραγκίσκος. Θα δουλεύουμε λιγότερο για να παράγουμε κάτι πλέον. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ξέρω ότι παράγουμε πολύ περισσότερα τρόφιμα με πολύ λιγότερα από ό,τι παλιά, με λιγότερο κόπο. Θα χρειαστεί μια προσαρμογή. Μέσο πρόθεσμα όμως. δεν νομίζω ότι θα υπάρχει λιγότερη απασχόληση. Βέβαια αυτό θα εξαρτηθεί από την ε, εξέλιξη των πραγμάτων. Επί παραδείγματι, εγώ προσωπικά από το που βγήκαν τα κινητά τηλέφωνα δουλεύω 24 ώρες το 24 ώρο. Παλιότερα οπωσδήποτε δουλεύα λιγότερο. Ε, θέλει κανείς να τοποθετηθεί στην πρόκληση αυτή του αυτοματισμού και της ψηφιοποίησης ως προς το ωράριο εργασίας του καθενός. Παρακαλώ εσείς. Εγώ το ανέφερα αυτό το θέμα ε, στην ε, παρουσίασή μου. Δεν είχατε καταφτάσει ακόμα. Και είναι μια ανησυχία που αφορά περισσότερο τις βιομηχανικές χώρες. Είναι ενδιαφέρουσα αυτή η διαδικασία όταν η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη ε, λαμβάνει διαρκώς όλο και περισσότερο χρηματοδότηση, ιδίως στις μεγάλες πόλεις. Αντιθέτως όμως υπάρχουν και αγροτικές περιοχές όπου βεβαίως η ψηφιοποίηση επίσης είναι πολύ σημαντική, αλλά όπου η οικονομία δυστυχώς συρρυκνώνεται. Πρόκειται για μια διαρκώς ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο στον, ε, στην αγορά εργασίας, στην οικονομία. Γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική η, η κατάσταση. Οι θέσεις που έχουμε εμείς είναι ότι προφανώς ορισμένες πτυχές της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης βεβαίως και μπορούν να αποφέρουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Άρα αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν αποτελεί μονοδιάστατα μια απειλή, αλλά είναι ανάγκη να βρούμε εκείνα τα αντισταθμίσματα στην αγορά εργασίας και να εξασφαλίσουμε και τους, τα επαγγέλματα που θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που απασχολούνται στην ε, παροχή φροντίδας, φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα, δεν εξαφανιστούν. Οι λύσεις πρέπει να είναι βιώσιμες και μακρόπνοες. Τα χρήματα που κατευθύνονται στον τομέα των ε, υπηρεσιών φροντίδας είναι πάρα πολύ ε, λίγα. πολλές φορές πέφτει στους ώμους των γυναικών, ε, των κοριτσιών να φροντίζουν τους ηλικιωμένους τους. Και πολλέ φορέ είναι και μια παροχή υπηρεσία η οποία δεν αναγνωρίζεται. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που αφορά την αγορά εργασία που πρέπει να εξεταστεί. Ξέρω ότι δεν έχω εγώ τώρα τη λύση να σας δώσω δυστυχώ. Ξέρω ότι πολλού του απασχολεί αυτή η ψηφιοποίηση. Νομίζω όμως μια απάντηση θα μπορούσε να είναι να οικοδομηθούν εταιρικέ σχέσεις, να γίνουν συνεργασίες, συμπράξεις, όπου θα υπάρχει ένας πραγματικός διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να εξα... εξεταστεί πραγματικά πώς μπορεί να διαμορφωθεί αυτό το μέλλον της Ευρώπης με επίκεντρο τον άνθρωπο και πώς μπορούν οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές οργανώσεις να συμβάλλουν σε μια τέτοια διαδικασία. Και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς στην κάρτας Ευρώπη ε, είναι πολύ αυτή η, αυτό το μοντέλο της κοινωνικής επιχειρηματικής επιχειρηματικότητας. Δεν είναι ακριβώς αυτό που αναφέρατε εσείς ως παράδειγμα από την Ισπανία, αλλά μιλούμε για επιχειρήσεις που ε, θα είναι μεν κερδοφόρες, θα είναι κερδοσκοπικές, αλλά αυτές, αυτά τα κέρδη που θα αποκομίζουν θα επιστρέφουν στην κοινωνία μέσω κοινωνικών επιχειρήσεων. Όπως για παράδειγμα υπάρχει το ξενοδοχείο Μάκτας στην Βιέννη. Ξενοδοχείο, πραγματικό, κανονικό, ε, το οποίο το, ε, το λειτουργούν πρόσφυγες οι οποίοι δεν θα είχαν διαφορετικά πρόσβαση στην αγορά εργασίας λόγω του νομικού καθεστώτος ε, στο οποίο εντάσσονται, εμπίπτουν αυτή τη στιγμή. Να ένα παράδειγμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε διάφορα τέτοια παραδείγματα, διάφορες τέτοιες ιδέες και στο πλαίσιο αυτό βεβαίως μπορεί να αξιοποιηθεί και η διαδικασία της ψηφιοποίησης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως υπάρχει ένα πρόβλημα, τουλάχιστον που αντιμετωπίζουμε εμείς στην Ελλάδα, σχετικά με το ωράριο εργασίας. Παραδείγματο χάρη, ο δημόσιο τομέα, που είναι ο κρατικό τομέα, εκεί το ωράριο τηρείται επακριβώ. Θα έλεγα μάλιστα πολλέ φορέ μειώνεται κιόλα. Στον ιδιωτικό τομέα όμω, με το φάσμα τη ανεργία και με την απειλή ότι θα χάσει την εργασία, έχει χαθεί το ωράριο. Ακόμη και σε επαγγέλματα που θεωρούνται πολύ αξιοπρεπή, όπως παραδείγματο χάρη του τραπεζικού υπαλλήλου, σήμερα στις τράπεζες, στις ιδιωτικές και εκεί ακόμη έχει χαθεί το ωράριο. Δηλαδή υπάρχει μια υπερπίεση εργασίας προκειμένου να μειωθεί το κόστος. Και φυσικά αυτό δημιουργεί όντω προβλήματα που έχουν να κάνουν στη συνέχεια με την ψυχολογία του ανθρώπου που εργάζεται, με την οικογένειά του και τον χρόνο που έχει απολέσει. Και εκεί έρχεται η Εκκλησία πολλές φορές όσο μπορέσει να δημιουργήσει ευκαιρίες, διότι πλέον ακόμη και η ψυχαγωγία κοστίζει. Άρα όταν δημιουργούμε προϋποθέσεις οι άνθρωποι να μπορέσουν να έχουν έναν χώρο ή έναν τρόπο να ξεκουραστούν και ψυχικά και σωματικά χωρίς υπερβολικό κόστος, αυτό είναι σήμερα μια κοινωνική προσφορά. Δεν ζητούν οι άνθρωποι πάντοτε μόνο ψωμί και φαγητό. Ζητούν και τρόπο να ζήσουν κάποια στιγμή απελευθερωμένοι από την πίεση που δέχονται πολλές φορές δυστυχώς στις σημερινές συνθήκες εργασίας. Ακόμη και επαγγέλματα που θεωρούνται πολύ πιο αξιοπρεπή στο παρελθόν είναι μια πραγματικότητα. Η Ελλάδα το ζει σε πιο έντονο, πιστεύω, χαρακτήρα και τρόπο, αλλά έχω την αίσθηση ότι ακόμη και σε άλλα μέρη της Ευρώπης συμβαίνουν παρόμοια παραδείγματα. Ναι, θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε... Ε, δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για εργασία ως μια δραστηριότητα. Είναι μια δραστηριότητα που πρέπει να πραγματοποιείται σε όρους ποσοτικούς τώρα, μέσα σε συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένα όρια χρονικά, προθεσμίες. Και θεωρώ ότι μπορεί να υπάρχει και σπάνιος εργατικού δυναμικού χωρίς να μπορώ να μιλήσω για όλη τη Βουλγαρία, αυτό το βλέπουμε κυρίως στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, τουλάχιστον δική μου την περιοχή. Υπάρχει σπάνιε εργατικού δυναμικού. Το Ισλάμ καλεί τον εργαζόμενο να βελτιώνει διαρκώ τι δεξιότητε και τι ικανότητε του. Ταυτόχρονα έχουμε για την, πολιτική, την κοινωνική πολιτική, γιατί δεν έχουν όλοι ούτε τους ε, ε, πνευματικούς σπόρους, το δυναμικό για να εξελιχθούν. Αν δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε σε όρους τεχνητούς ε, απασχόληση, ίσως θα μπορούσαν να δεχθούν μια λιγότερο ε, καλή αμοιβή για μια πιο τετριμένη επαναληπτική εργασία. Χωρίς αυτό να είναι στόχος, θα ήταν ίσως σκόπιμο στην κοινωνική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να προβλέψουν για όλους εκείνους οι οποίοι δεν είναι προνομιούχοι, είναι λιγότερο μπροστά στην αγορά εργασίας, γιατί και σε αυτούς πρέπει να δώσουμε προσοχή. Αλλιώς θα βρεθούν σε ανταγωνιστική τα κράτη μεταξύ τους και με, τους, ε, με τον έξω ανταγωνισμό. Ο πρόεδρος... Να... αγγλικά λοιπόν για να γίνουμε πιο οικουμενικοί. Ε, πολλά ήταν τα ενδιαφέροντα που υπόθηκαν, αλλά ιδιαίτερα θέλω να φερθώ στα όσα είπε ο Σεβασμιότατο Ιγνάσιο. ότι, ότι δηλαδή όταν κανεί βρίσκεται στη θέση που μπορεί να εκβιάσει, να πει «Α, θα κάνεις αυτό που θα σου πω». Καταχρηστικά. Ιδάλλως θα χάσει τη δουλειά σου. Δεν υπάρχει καμία έννοια αξιοπρέπειας Εκεί ο έλεγχος, ο νόμος, ο έλεγχος του νόμου, η εφαρμογή του νόμου πρέπει να παρεμβαίνει. Αυτά που μπορούν να έρθουν με τη νέα τεχνολογία μπορούν να φέρουν και αυτό το δεδομένο. Και θα απαντήσω στα ισπανικά ότι είναι δύσκολο να φανταστούμε το μέλλον, ιδιαίτερα σε αυτή τη μεταβατική περίοδο φαίνεται ότι, είναι, ότι είμαστε καταδικασμένοι, ότι είναι αναπόδραστο αυτό το μέλλον. Τα πράγματα βαίνουν πολύ γρήγορα. Χρειάζεται όμως ο άνθρωπος περισσότερο χρόνο, περισσότερο χρόνο για να βρει τον τρόπο να προσαρμοστεί και θα, γι' αυτό θα χρειαστούν νέες δυνατότητες για απασχόληση και πάλι με ισορροπία. Ίσως ε, σε όρους μελέτης ε, νέων σπουδών κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος όταν, όταν θα μείνει ελεύθερος χρόνος θα θελήσει να βρει κάτι να τον γεμίσει. Και θα πρέπει πάλι να σωσκελιστεί ο χρόνος απασχόλησης και μεταξύ των εργαζομένων. Βεβαίως μια νέα κατανομή του κεφαλαίου και περισσότερα κοινωνικά χαρακτηριστικά του κεφαλαίου, όπως με τις συνεταιριστικές οργανώσεις, μπορεί να είναι οπωσδήποτε μια πολύ σημαντική λύση. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται χρόνος. Βρισκόμαστε στην επαρχή μιας επανάστασης σε εποχές δύσκολης προσαρμογής, αυτή είναι η γνώμη μου. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί όντως αυτή η προσαρμογή είναι προσαρμογή που όλοι πρέπει να αναλάβουμε και εσείς με την προσαρμογή των πολιτικών ή των θρησκευτικών ε, θέσεων γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη αλλά αυτή η προσαρμογή δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της αξιοπρέπειας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία κάθε παρέμβαση. Άλλες ερωτήσεις παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ. τι ονομάζομαι. Από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γυναικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εξαιρετικές σας ε, παρουσιάσεις. Μια μεγάλη ανησυχία για μένα είναι το γεγονός ότι στο οικονομικό σύστημα το άτομο βρίσκεται στην καρδιά της ανάπτυξης της οικονομίας. Ενώ στις θρησκείες δεν έχουμε στο επίκεντρο, στο επίκεντρο το άτομο, αλλά το κοινωνικό σύστημα, το άτομο μεν, αλλά μαζί με τον οικογενειακό του περίγυρο, τους αγαπημένους του ανθρώπους. Αυτή είναι το, το, η καρδιά αυτών των συστημάτων. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρωτοβουλία ε, που έχετε αναλάβει. Ε, για, για τον ε, διάλογο και τη διαβούλευση με τις ε, θρησκείες, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το κοινωνικό περιβάλλον στην Ευρώπη. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε πώς η οικονομία μπορεί να καταστεί πιο υγιής, μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου ως πιστή ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας σύγκρουσης γιατί υπάρχει αυτή η αντίφαση ανάμεσα στο άτομο ως επίκεντρο της οικονομίας και της οικογένειας ως επίκεντρο της, της θρησκείας, της θρησκευτικής ζωής, της πνευματικής ζωής. Πώς μπορούμε, ε, σεβασμιότητε, ε, ε, γνάτη είπατε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, μήπως μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα, ποιες, είναι οι δικές σας θέσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώ έχει δοθεί η αίσθηση ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να σώσουν μόνο το άτομο. Και έχει χαθεί αυτό που εμείς ονομάζουμε στη δική μας παράδοση κοινότητα. Μια κοινότητα που υπενήχθη ο κύριος Πρόεδρος όταν μιλούσε για μοναστήρια. Βεβαίως δεν θα μιλήσουμε εδώ για τα μοναστήρια, αλλά εντούτοις τα μοναστήρια κατόρθωσαν να έχουν μια κοινωνική διαβίωση όπου υπερβαίνει τις δυνατότητες να χαθεί ένας άνθρωπος και σώζονται όλοι μαζί. Θα σας φέρω όμως ένα παράδειγμα από τη δική μου δικαιοδοσία. Είμαι σε μια περιοχή όπου ζούμε 250.000 άνθρωποι. Έχουμε περίπου 150 ενορίες, μικρές και μεγάλες, σε δύο πόλεις και χωριά. Και αυτή τη στιγμή εθελοντές, γυναίκες ως επιτοπλίστων, παράγουν κάθε μέρα 2.000 μερίδες φαγητό για ανθρώπους που δεν μπορούν να έχουν το φαγητό της ημέρας και παίρνουν ζεστό φαγητό κάθε μέρα. Όλα τα χρόνια τώρα πλέον. Στην αρχή όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα ήταν για συνήθως μη Έλληνες, πρόσφυγες, φιλοξενουμένους. Σήμερα είναι για Έλληνες. Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει καμία επιχορήγηση. Δεν τη χρειάζεται. Πολλές φορές οι ίδιες οι γυναίκες που μαγειρεύουν φέρνουν και τα φαγητά που θα μαγειρέψουν για τους άλλους. Πιστέψτε με ότι εμένα με ενδιαφέρει όχι μόνο αν θα πάνε φαγητό αυτοί που δεν έχουν, οι γυναίκε που μαγειρεύουν, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωφέλεια νιώθουν. Αυτό είναι έργο εκκλησίας, είναι έργο κοινότητα. Καταλαβαίνω ότι ανήκουν σε μια ευρύτερη οικογένεια που λέγεται ενορία. Και αυτό βοηθάει ψυχολογικά, ψυχικά, σώζει πέρα από το θρησκευτικό. Πιστεύω ότι δυστυχώ η Ευρώπη πολλέ φορέ χάνει αυτή την κοινότητα. Προσπαθεί να δημιουργήσει άλλε δομέ, αλλά οι εμπειρίε δεν είναι οι καλύτερε από τι άλλε δομέ. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Σας λέω αυτό που ζούμε εμείς. Και αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την κρίσιμη περίοδο και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή την αίσθηση ότι έχουμε και μία ενοποιό δύναμη που λέγεται πίστη. Αυτός που πιστεύει αντλεί δύναμη την ώρα που το έχει ανάγκη και δεν περιμένει μόνο από τις υλικές απολαβές. Και έρχεται μετά και η ώρα που θα ξεπεράσουμε, ελπίζω, και τα οικονομικά προβλήματα. Σας ευχαριστώ. On s'excite. Ανάβουν τα αίματα, αλλά δεν έχουμε πια τόσο πολύ χρόνο. Κύριε Πυρίνσκι, ζητήσατε εσεί το λόγο. Κύριε Πυρίνσκι, όχι. Α, λάθο έκανα. Μία, δύο, τρει. Και σταματούμε αν έχετε την καλοσύνη, εκτό και αν η πρόεδρο θέλει να συνεχίσει. Ακόμη ένα. Αλλά δεν βλέπω gender balance, δεν βλέπω ισότιμη εκπροσώπηση των φίλων. Τέλο πάντων, να κλείσουμε το με του τέσσερι. Γιατί με περιορίζει και η, η δική μου η ατζέντα έχω εδώ, το χωροφύλακα που θα με σταματήσει δίπλα. Παρακαλώ, κύριε Τσάμπον. Θα μιλήσω αγγλικά εκ μέρους της Βρετανικής Κοσμικής εταιρεία στη μη θρησκευτική δηλαδή πλευρά του διαλόγου. Θέλω να, ζητήσω μια, να κάνω μια έκκληση για την αξιοπρέπεια εκείνων που ζητούν ισότητα και αξιοκρατία. Όλο και περισσότερο μαθαίνουμε, ε, έχουμε πληροφορίες ε, για δασκάλους θρησκευτικών σε σχολεία δημόσια, με δημόσια δηλαδή χρηματοδότηση, που απολύονται επειδή δεν έχουν τη θρησκευτική πίστη, ε, μάλλον στα θρησκευτικά σχολεία, αλλά δεν διδάσκουν θρησκευτικά, και επειδή έχουν χάσει τη θρησκευτική πίστη, αυτοί απολύονται. Δηλαδή, πόσο πρέπει να είναι κανεί θρήσκο, γιατί πρέπει να είναι κανεί θρήσκο για να διδάξει μαθηματικά, φυσική ιστορία. Είναι δυνατόν να απαιτείται να ακολουθεί κανείς το θρησκευτικό, τη θρησκευτική πίστη. Ε, δεν πρέπει να, αρχούν, να αρκεί η αξιοκριτία, ο καλύτερος δηλαδή και ικανότερος να προσλαμβάνεται. Και θα ήθελα προχωρώντας να αναφερθώ στο γενικότερο ζήτημα του κοινωνικού πυλώνα με μεγαλύτερη θρησκευτική συμμετοχή που αναφέρθηκε. Νομίζω ότι ο κίνδυνος θα ήταν να ενισχυθεί η παρουσία της θρησκευτική διάστασης στην Ευρώπη και να αισθανθούν εκείνοι οι οποίοι δεν ανήκουν σε μια θρησκεία ε, πως είναι στο περιθώριο. Ιδιαίτερα εκείνοι που είναι ομοφιλόφιλοι, που δεν έχουν οικογένεια ή δεν έχουν ε, παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο, να αισθάνονται ότι αποκλείονται από, την, από τον διάλογο αυτόν. Αυτή είναι η έκκλησή μου και σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Έχω λίγα εγώ να σχολιάσω εδώ. Μόνο συνεχίστε τον αγώνα και είμαστε στο πλευρό σας. Γιατί είναι και αυτές αξίες της Ευρώπης. Δεν ξέρω εάν ε, οι προσκεκλημένοι μας, παρακαλώ. Πώς θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να παρατηρήσω ότι φαινόμενα όπως τα περιγράψατε δεν έχουν να κάνουν καθόλου με την Ελλάδα τουλάχιστον. Εκεί είμαστε καλά Κανείς δεν χάνει την εργασία του εξαιτία του αν πιστεύει ή δεν πιστεύει στην Ελλάδα και σε κανένα χώρο. Αυτό όμω που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι το δικό μας μήνυμα είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, όποιο και αν είναι, από όπου και αν προέρχεται, ό,τι και αν πιστεύει, είναι μια ζωντανή εικόνα του Θεού. Και εμείς αυτό κηρύττουμε. Και όπω όταν έχουμε, εμεί ξέρετε, οι Ορθόδοξοι τις εικόνες που τι σεβόμαστε πάρα πολύ, τι αγαπάμε, τι έχουμε σαν θησαυρό, αν αυτό αφορά ένα αντικείμενο που είναι φτιαγμένο με ανθρώπινα χέρια, καταλαβαίνετε πώς αγαπάμε τον κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι το κηρύγμά μας. Ίσως δεν το εκφράζουμε σωστά στην πράξη πάντοτε. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι αν παραμείνει αυτό το κήρυγμα στους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν, τότε οι όποιοι άνθρωποι ακόμη και αν δεν πιστεύουν θα νιώθουν και ελεύθεροι και θα ζουν και με αξιοπρέπεια, γιατί θα τους στηρίζουν οι άνθρωποι της πίστεως. отношение на назначаването на, на човек... Όσον αφορά την ε, επιλογή κάποιου σε μια θέση, το Ισλάμ μας λέει ότι πρέπει να επιλέγουμε τον καλύτερο. Απλώς λέει ότι ο πιστός Εάν έχει ανάγκη από 5-10 λεπτά για την προσοχή του μέσα στο ώρο, δεν χρειάζεται να αποχωρήσει από το χώρο εργασίας του και πρέπει να αναζητήσει τον, ε, την ισορροπία ανάμεσα στην, στον προσωπικό και τον επαγγελματικό βίο. Είναι οπωσδήποτε πολύ εύκολο εάν το θέλει και ο εργοδότης να διευκολύνει. Hablaré en español. I speak Spanish. <clears throat> Ένα σχόλιο θα ήθελα να κάνω και μετά μια ερώτηση. Όσον αφορά τον ε, συνδυασμό επαγγελματική και προσωπική ζωής, εμεί έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία χριστιανοί, καθολικοί και Προτεστάντε, που είναι με τίτλο «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Κυριακή». Ε, αφορά και την ψηφιοποίηση. Κάποιοι το προσεγγίζουν από, από, τη σκοπιά ε, της πίστης, άλλοι όχι. Η Σάνων μίλησε για την νεολαία και αντιμετωπίζουμε μια σειρά από προβλήματα, ιδιαίτερα στο Νότο, στην Ισπανία. Αυτό που είπατε, η φυγή εγκεφάλων, η ανεργία, Και πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο συνδέεται βεβαίως με τα κοινωνικά δικαιώματα αλλά και με την έλλειψη συμμετοχής. Η Καθολική Εκκλησία πρόσφατα για πρώτη φορά ε, διοργάνωσε μια συνδιάσκεψη με νέους ανθρώπους για να τους ρωτήσει, για να ακουστεί η φωνή τους. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και από τους άλλους εκπροσώπους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, το Ισλάμ, τι μέτρα έχουν πάρει για τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δυστυχώς εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχουμε τον τρόπο της Καθολικής Εκκλησίας να συγκεντρώνουμε όλους τους νέους από όλο τον κόσμο. Λειτουργούμε ως επιμέρους τοπικές εκκλησίες έχοντας την ενότητα της πίστεως αλλά αναλαμβάνοντα την ευθύνη των νέων τη κάθε περιοχή ο επίσκοπό του ω επιτοπλίστων. Και βεβαίω εκεί εξαρτάται από του θεσμού που δημιουργούνται. Δεν είμαστε τόσο όσο θα θέλαμε ευχαριστημένοι στο διάλογο με του νέου. Είμαι απόλυτα ειλικρινή μαζί σα. Όμω τον αναζητούμε, το προσπαθούμε. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματο χάρη στην περιοχή μου, όπου έχουμε κατασκηνώσει για νέου το καλοκαίρι, είμαστε υποχρεωμένοι να αρνηθούμε αιτήσει γιατί δεν έχουμε χώρο δεν μπορείτε δεν να φανταστείτε πόσο μας δυσκόλεψαν οι νότες της Ευρώπης στο να κάνουμε τις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων. Μας αντιμετωπίζουν τις κατασκηνώσεις της Εκκλησίας ως να είναι ιδιωτικέ που βγάζουν χρήματα. Να μέσα μέσα ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε τις νότες που θέλουν όντως να διασφαλίσουν, απ' την άλλη όμως ένας ιδιώτης που είναι επιχειρηματίας έχει τον τρόπο. Θα σας φέρω το πιο απλό παράδειγμα. Να έχει του χάρη οπωσδήποτε ένα γιατρό στην κατασκήνωση κάθε μέρα. Ε, Εμεί δεν μπορούμε αυτό εύκολα να το κάνουμε γιατί δεν υπάρχει γιατρό που να αφήσει το ιατρείο του και να έρθει στην κατασκήνωση. Βλέπετε λοιπόν αμέσω αμέσως ότι υπάρχουν θέματα. Εν τούτης, εμείς χαιρόμαστε την ευρωπαϊκή παρέμβαση στην ασφάλεια των παιδιών και στο ΣΥΤ λειτουργία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να απαντήσω τελικά, προσπαθούμε και εμείς το διάλογο αυτό, να φέρουμε τη φωνή των νέων μέσα στην Εκκλησία και το κάνουμε με όποιο τρόπο μπορούμε κάθε φορά καλύτερο. Ευχηθείτε να κάνουμε ακόμη κάτι πιο πολύ. младостта от гледна точка на исляма, предполагам от всички. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πλούτος είναι για το Ισλάμ, είναι το μέλλον μας, είναι αυτό που μας, έχει, μας ε, εξασφαλίζει το μέλλον. Κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να συνεργαστούμε μαζί τους, με τους νέους, με τις οικογένειες. Προσπαθούμε να έχουμε τακτική επικοινωνία μαζί τους. Ιδιαίτερα λοιπόν λέει στο νέο η θρησκεία μας διάβαζε, ε, απόκτησε γνώση άνοιξε τα μάτια σε όλη την κοινωνία και επιδιώκουμε να υπάρξει μια πραγματική εξέλιξη με επικοινωνία με τους νέους, σε επικοινωνία με τους νέους. Και βέβαια σε αναζήτηση και του χρόνου που χρειάζεται για να τα καταφέρουμε όλα αυτά, γιατί δεν είναι τίποτε παγιωμένο ή χαραγμένο σε μάρμαρο. Παρακαλώ. Άλμπερ Γκίγκη, Μέγα Ραβίνο των Βρυξελών. Ξεκινώντα, θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Μαγκίνο, πρώτη αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που μα επέτρεψε να συνευρεθούμε γύρω από το θέμα αυτό που είναι άκρο σημαντικό όσο και περίπλοκο. Περίπλοκο γιατί δεν ξέρω προς τα πού πρέπει να κινηθούμε, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε για να αναστήσουμε τη λύση όλο και περισσότερο σήμερα. Βλέπουμε αυτό που έχει σημασία στην κοινωνία μας να είναι η αποδοτικότητα. Μόλις πέσει η αξία των μετοχών, αμέσως καταδικάζεται ο εργαζόμενος, ο εργάτης. Εταιρείε μπορεί να βγάλουν χιλιάδες εργαζομένων στην ανεργία επειδή μειώθηκε η αποδοτικότητά τους η παραγωγικότητα. Επομένως, δεν ε, εγγράφεται πλέον στο επίκεντρο της οικονομίας του ανθρώπινο αλλά η οικονομία έχει καταλάβει την κυρίαρχη θέση παντού. Δεν ξέρω πώς μπορούμε αυτό να το αντιπαλέψουμε. Γιατί είναι ένα πρόβλημα. Ωστόσο, με ε, εξέπληξε η μαρτυρία του Μητροπολίτη Ιγνάτιου, του Ιγνάτιου και θα ήθελα να κάνω μια πρόταση που νομίζω δεν θα είναι δύσκολο να υλοποιηθεί και θα κοστίσει και πολλά. Ξέρουμε ότι σήμερα όσοι έχουν ε, γνώσεις και δεξιότητες εργάζονται ως τα 65 τους, ότι η διάρκεια ζωής είναι όλο και μεγαλύτερη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ικανότητες, έχουν δεξιότητες, θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν, να προσφέρουν. Και είναι νομίζω πολύ σημαντικό σήμερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλιστεί ένα καθεστώς των εθελοντών. Μπορούμε να δώσουμε, πρέπει να δώσουμε μία θέση στους εθελοντές, ώστε να μην αισθάνονται παρήσακτοι. Διότι σήμερα όταν πάνε κάπου ε, τους κοιτάνε με δυσπιστία, με φόβο, λένε «Α, θα έρθει να μου πάρει τη θέση εμένα που έχω τη δουλειά αυτή» κτλ. Μα έχουμε τόση μεγάλη ανάγκη αυτών των εθελοντών στις κοινωνίες μας που έχουν ικανότητες και γνώσεις καταπληκτικές και που ένα μόνο ζητούν να τους επιτραπεί να δώσουν, να προσφέρουν και μόνο να προσφέρουν γιατί ξέρουν ότι όταν προσφέρουν λαμβάνουν. Έχουμε τι διοικητικέ υπηρεσίε που μπορεί να χρειάζονται για προσωπικότητα, νοσοκομεία, τι βιβλιοθήκε. Όλα αυτά, αλλά πρέπει να του αναγνωριστεί ένα καθεστώ με το ρόλο του, ε, του εθελοντή, ώστε να μην αισθάνεται παρήσακτο ή περιθωριακό, ότι ίσα ίσα τον ανέχονται με τα βία. Όχι, να βρει τη θέση του την πραγματική. Και είναι πολύ σημαντικό. Και θα βοηθήσει σε όρους εκθετικούς την κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ το Μαγαραβινό. Την τελευταία στιγμή αυτού του κομματιού της συζήτηση μας βγάζεται ένα τόσο σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα. Ε, θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η πλάστιγκα, έχω λιγότερη δουλειά γιατί προχωρεί η ψηφιακή τεχνολογία τη δουλειά που μας μένει, μας την ε, τρώνε οι εθελοντές. Ε, όχι, σας καταλαβαίνω απολύτως, εγώ είμαι υπέρ της εθελοντικής εργασίας. Είμαι μάλιστα και σκιώδης εισηγητής μιας πρότασης πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σώμα αλληλεγγύης που ε, ευνοεί την αναγνώριση. Σαν αστείο το είπα αυτό με την πλάστιγκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή τις θέσεις και του ρόλου του εθελοντή, γιατί έχετε δίκιο, παρότι προσφέρουν τόσα πολλά και καλά στην κοινωνία, δεν ε, την χάνουν βοήθειες. Δεν θέλω να προχωρήσω στη συζήτηση αυτή τώρα, αλλά θα έχετε εσεί την ευκαιρία, φαντάζομαι, να επανέλθετε. Ένα κύριο και μια κυρία. Α αφήσω την κυρία τελευταία για να μην με κατηγορήσει κανεί ε, για ζητήματα ισότητα ε, στην εκπροσώπηση των φίλων. Παρακαλώ εσεί. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε στη συζήτηση ότι στην αγορά κυριαρχεί η επιλογή του κεφαλαίου και ο Σεβασμιότατος χρησιμοποίησε τον όρο μισθή ε, φτώχειας, μισθή μιζέριας, έχει μεταφραστεί αυτό στα γαλλικά. Ε, μήπως λοιπόν πρέπει να συνδεθεί αυτό το θέμα με την αξιοπρέπεια του μισθωτού και του εργαζομένου. Ε, έτσι θα δώσω ένα παράδειγμα στα λογιστικά συστήματα που έχουν σε κάθε επίπεδο οι επιχειρήσεις και, στα, και οι πολυεθνικές ακόμη, τον μισθό τον ε, καταγράφουν ως κόστος. Δηλαδή κάθε φορά που έχουμε πρόβλημα οικονομικό πρέπει να μειωθεί το κόστος, δηλαδή ο μισθός. Από την άλλη, τα κέρδη και ωφέλη θεωρούνται ως κάτι πολύ καλό, μου πρέπει να ξαναδιανεμηθεί στον μέτοχο και μόνο στους μετόχους, στον μέτοχο στους μετόχους. Μήπως λοιπόν εκεί θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί και να προσπαθήσει να εξετάσει αυτά τα λογιστικά συστήματα που έχουν πλέον θεσπιστεί ε, από τις μεγάλες πλέον τράπεζες, μεγάλες πολυεθνικές και που έχει δεχθεί χωρίς ε, καν, να αντιδράσει το παραμικρό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως είναι αυτό μια ευκαιρία να αντιστρέψουμε το ζήτημα και το τον προβληματισμό της αξιοπρέπειας στον χώρο εργασίας. Επίσης έχουν γίνει πολλές μελέτες που αποδεικνύουν ότι μεγάλες πολυεθνικές και κυρίως στις ε, ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κάνουν σεβαστό το χάρτη των θεμελιωδών ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ρωτώ λοιπόν, δεν πρέπει κάτι να γίνει σε αυτό, ώστε να επιβληθεί σε αυτές τις ε, μεγάλες εταιρείες να κάνουν σεβαστό τουλάχιστον, τουλάχιστον το χάρτη των, των θεμελιωδών ελευθερών και δημοκαιωμάτων. Γιατί αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για το σεβασμό της αξιοπρέπειας. Με συγχωρείτε, δεν συστήθηκα από την ε, Ένωση ΕΓΚΑΛ, Ισότητα, Ευρώπη και Κοσμικότητα, ε, άρα εκπροσωπώ την κοσμική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θέτεται ένα ενδιαφέρον ζήτημα προς συζήτηση. Δεν θα έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε, αλλά έχουμε εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, οι οποίοι καταγράφουν τις ε, προτάσεις και ιδέες σας. Πάντως το Κοινοβούλιο ε, ασχολείται ιδιαίτερα με, τις, με τα λογιστικά πρότυπα, πρότυπα, σε όρους τεχνικούς ίσως, όχι τόσο ηθικούς, αλλά... Πιο πολύ δεν μπορούμε να το αναλύσουμε αυτή τη στιγμή, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο και η κυρία για να ολοκληρώσουμε. Τι αρκεία από το Religion for Peace και του WCRP μέσα στο Religion for Peace. Έχουμε νέους Ορθόδοξους, Μουσουλμάνους, Εβραίους, δύο, από δύο Καθολικούς 25 χρόνια ασχολούμαι με τους νέους ε, στις κοινωνίες, στις κοινότητες που ζουν και έχω προσπαθήσει να τους αγκαλιάσω. Για το Εφτάρ, την θρησκευτική ε, γιορτή κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού όπου σταματάει η νηστεία. Ε, προσπαθούμε να ε, φέρνουμε μαζί τους νέους, να πηγαίνουν επισκέπτονται τους άλλους που το γιορτάζουν. Είναι μια ευκαιρία για να ε, γνωριστούν. Ήταν για τους εκπροσώπους μας της Χάιφα που πήγαν στην Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Τα γνωρίζουν αυτά. Το μόνο που χρειάζονται είναι υποστήριξη από το κράτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ και έτσι κλείνουμε με μερικά λόγια για τους νέους. Πάρα πολύ ωραία. Μετά αυτές τις σκέψεις θα δώσω σύντομα το λόγο στον ε, σεβασμιότατο Ιγνάσιο και Ιγνάτιο και στον Μουφτή και την κυρία Φόμαν για να ολοκληρωθεί ε, η συζήτηση με τα συμπεράσματά τους. Εγώ δεν έχω τίποτε άλλο να προσφέρω, να συμπληρώσω παρά μόνο ότι ευχαριστώ θερμά για τη δυνατότητα που είχα να λάβω μέρος σε αυτή την τόσο σημαντική συνάντηση. Ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο κυρία Μαγκίνες. Αφήνω τη θέση για να την καταλάβουν οι επόμενοι, αλλά πρώτα απ' όλα εσείς αν θέλετε σεβασμιότατε, αν θέλετε να λάβετε το λόγο, κυρία δώσατε να είμαι ανάμεσά σας. Ομολογώ ότι είναι η πρώτη μου εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ θετική εμπειρία. Εύχομαι να συνεχίσετε, κυρία Πρόεδρε, με τον ίδιο πόθο και τρόπο να συζητάτε και με αυτούς που εκπροσωπούν την πίστη και τη θρησκεία και με αυτούς που είναι απέναντι στην πίστη και στη θρησκεία. Ο διάλογος θα δώσει την αλήθεια και η Ευρώπη πρέπει να κρατήσει αυτή τη μεγάλη αξία του διαλόγου σε ό,τι αφορά την παρουσία μου, επιτρέψτε μου να την αφιερώσω στα πιο αγαπητά παιδιά που έχω εκεί στην πόλη που ζω, στο Βόλο, στα Ρωμά παιδιά, με τα οποία με αθλητισμό, με ένα μικρό πρόγραμμα που πήραμε και με κάθε τρόπο που προσπαθούμε να κάνουμε για να τα έχουμε ενταγμένα μέσα στην κοινωνία μας, έχουμε πετύχει κάτι που δεν γίνεται με άλλες δομές, αλλά μόνο με τους εθελοντές και ευχαριστώ το Ραβίνο που έθεσε το θέμα. Το χρειαζόμαστε το πρόβλημα και το θέμα των εθελοντών, διότι λειτουργούμε πολλές φορές μεταξύ παρανομίας και νομιμότητας. Εγώ όμως αφιερώνω στα Ρωμά παιδιά μου αυτή τη συνάντηση και σας ευχαριστώ πολύ. За мен също е огромна чест днес да бъда участник в този висок форум. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν και για μένα πολύ μεγάλη η τιμή που μπόρεσα να συμμετάσχω σε αυτό το φόρουμ υψηλού επίπεδου. Οπωσδήποτε και προφανώς ε, η αξιοπρέπεια του εργαζομένου ξεπερνά την ε, απλή εργασία που παράγει, το απλό έργο που παράγει. Επιτρέπει δηλαδή στον άνθρωπο να αναπτύξει την προσωπικότητά του. Ο εργαζόμενος δεν πρέπει απαραίτητα να έχει αναλάβει ένα έργο πολύ περίπλοκο στην θρησκεία μας στο Ισλάμ. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η καλή ανατροφή, η καλή εκπαίδευση, χάρη στην οποία, η παιδεία ούτως επίν, χάρη στην οποία μπορεί κανείς να βρει και μια θέση εργασίας αργότερα. Ο άνθρωπος, εκείνος που εργάζεται, είναι ένας πλούτος για την κοινωνία, είναι σημαντικός πόρος για την κοινωνία, όπως και για την επιχείρηση άλλωστε. Χωρίς τον ε, εργαζόμενο δεν θα είχαμε τίποτα να προσφέρουμε, δεν θα είχαμε τίποτα να παραγάγουμε. Και γι' αυτό πρέπει να ενισχυθεί η σημασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε κοινωνικό επίπεδο. Πρέπει να το εξασφαλίσει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φόμαν. Νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η στιγμή για να υπενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της πόσο σημαντικό είναι να ηγηθούν μιας διαδικασίας εξασφάλισης της ευημερίας για όλους, ότι δεν μπορεί στόχος να είναι μόνο το κέρδος, αλλά πρέπει να αναπτυχθεί ολόκληρη η κοινωνία συμπεριλαμβανομένων όλων των πολιτών της. Χρειάζεται προστασία των εργαζομένων από τη μία μεριά και ε, καινοτομία στην οικονομία. Πρόκειται για στόχους οι οποίοι συμβαδίζουν και δεν είναι καθόλου αντιφατικοί. Στη βάση αυτών καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, ενισχύσει τις προσπάθειές της ε, στον τομέα της κοινωνικής ε, επιχειρηματικότητας που συνδυάζει την ιδιωτική οικονομία με την κοινωνική αλληλεγγύη. Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων αποτελεί σημαντικότατο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μετουσιώσει το συντομότερο δυνατό σε συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις της διακηρύξης της μέσω του ε, Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Πρόεδρος, Πραγματικά ήταν εξαιρετικό το κλείσιμό σας και εγώ μπορώ να σας πω ότι συμμερίζομαι πλήρως ε, ως εισηγητής ε, για το θέμα της προβλεψιμότητας των εργασιακών σχέσεων ε, και στόχος μου πραγματικά είναι να εξασφαλίσουμε στην ολότητά της την αξιοπρέπεια των ανθρώπων στον χώρο εργασίας σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ λοιπόν για την παρουσία σας, για τις παρουσίες σας, για τη συμμετοχή σας, τη συμβολή σας. Σας εύχομαι ε, ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. And, and may I sincerely... Και να σας ευχαριστήσω εγώ κύριε Σαμπον γιατί νομίζω ότι έγινε εξαιρετική, εξαιρετικά ζωντανή η συζήτηση χάρη σε εσάς. Ε, και λόγω του κλεισίματος των καταληκτικών σας παρουσιάσεων, γιατί ως εισηγητής και μέλος της ε, Επιτροπής Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πραγματικά πιστεύω ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε τα όσα ακούστηκαν εδώ στη δουλειά σας σήμερα. Να ζητήσω από τους ομιλητές μας να κατέβουν κάτω στις, ε, στα έδρανά τους, σας παρακαλώ, για να έρθουν οι νέοι ομιλητές, οι ομιλητές του δεύτερου γύρου, να σας εξηγήσω πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα στο επόμενο πάνελ που, είναι, ε, που έχει τίτλο «Ενίσχυση και προώθηση μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας που θα συμπεριλαμβάνει όλα τα μέλη της και θα νοιάζεται». Καλωσορίζω τον συνάδελφό μου, τον κύριο Πυρίνσκι, που επίσης είναι μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και θα συντονίσει τη συζήτηση αυτή, ο οποίος και θα παρουσιάσει τους ε, ε, επόμενους ομιλητές μας. Ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, να σας, μου επιτρέψετε να σας πω, που ήταν γεωργός, έλεγε ότι η εργασία είναι προσευχή. Λαμποράρε ετοράρε, νομίζω είναι η αντίστοιχη έκφραση στα λατινικά και νομίζω ότι αυτό αποτελεί και την ουσία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Οι άνθρωποι χρειάζονται ένα νόημα στη ζωή τους, ένα, ε, ένα, μια οδό ε, για να μπορούν να προσφέρουν. Και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κανείς να είναι πάντοτε γονατιστός και να προσκυνά ή να προσεύχεται στο Θεό, αλλά να μπορεί πραγματικά μέσα στην καθημερινότητά του να προσφέρει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ε, είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε εξαιρετικά στο συντονισμό της από εδώ και πέρα συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Πυρίνσκι. Με πολύ μεγάλη μου χαρά προεδρεύω αυτού του γύρου συζητήσεων είναι δύσκολο το έργο αυτό βεβαίως, ε, ιδίως αφού διαδέχομαι τον κύριο Σαμπον με αυτήν την εξαιρετικά ζωντανή του παρουσία. Αυτό το πάνελ έχει τίτλο του «Ενίσχυση και προώθηση μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας που, χωρίς αποκλεισμούς που θα νοιάζεται και θα φροντίζει τα μέλη της». Ε, έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας ε, βάσει του χρόνου διαγράμματος που έχει καταρτιστεί έως τις 6 ε, αν δεν κάνω λάθος. Και θα πρότεινα να αξιοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας για να συνεχιστεί ο διάλογος αυτός, η συζήτηση αυτή που ήδη ξεκίνησε βεβαίως Μεταξύ άλλων θα πρότεινα να προχωρήσουμε γρήγορα γιατί υπάρχει και ένα όριο μέχρι το οποίο θα μας ε, ακολουθήσουν και θα μας συνοδεύσουν οι διερμηνείς. Ε, αν και νομίζω ότι εντάξει θα τα, θα τα καταφέρουμε. Ε, βλέπω ότι για εμένα είχαν προβλεφθεί περίπου 10 λεπτά. Απλά θέλω ούτε 5 λεπτά. Δύο-τρία πράγματα θα πω. Το πρώτο αφορά τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Δεν ξέρω βεβαίως σε ποιο βαθμό έχετε παρακολουθήσει το έργο αυτό εσείς ε, την ε, προσαρμογή και τη μετουσίαση σε πράξη αυτού του πυλώνα, αλλά είναι πραγματικά αξιέπαινο το γεγονός ότι προτάθηκε ο κοινωνικός αυτός πυλώνας από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προσπάθεια να ενισχυθεί πραγματικά αυτή η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ήταν διάχυτη η αίσθηση και είναι και προφανές ε, σε καθημερινό επίπεδο ότι ειδικά και ιδίω αυτή η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης αλλά και των τεχνολογικών εξελίξεων έχει αποδυναμωθεί στην λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων στα, κράτη-μέλη. Φιλοδοξία λοιπόν του Προέδρου Γιούγκερ ήταν να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κοινωνική με τριπλό α όπως, ε, ε, όπως αναφέρεται στα χρηματοπιστωτικά. Υπήρξε ε, έντονη συζήτηση. Κάποιοι είχαν προτείνει να υπάρχει ένα δεσμευτικό κείμενο το οποίο θα είναι θεσμοθετημένο και θα υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Στο τέλος αυτό στο οποίο καταλήξαμε είναι αυτό το άρθρο 12 του προημίου που λειτουργεί ως ε, κατευθυντήρια γραμμή για την επίτευξη αποτελεσματικής αποδοτικής εργασίας και την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις τις οποίες βεβαίως γνωρίζουμε όλοι και που εκτείνονται από τη διαδικασία της ψηφιοποίησης μέχρι την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής προσφυγικής κρίσης. Θα ήθελα να πω και εγώ αυτό που ανέφερε και η εκπρόσωπος της Κάρετας στις συνθήκες. Στη συνθήκη, για παράδειγμα, στο άρθρο 3 της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατοχυρώνεται ότι ε, ε, κατοχυρώνεται η έννοια της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς με πλήρη απασχόληση που θα εξασφαλίζει εδαφική και κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Ο πυλώνας λοιπόν με τη μορφή που έλαβε έρχεται να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το καθήκον, σε αυτή τη δέσμευση, δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθεί και να ενισχύει αυτή τη διάσταση της οικονομίας και της κοινωνίας. Να συνδυαστεί δηλαδή η, ο, η ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική ισότητα. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι ποια θα είναι η αλληλεπίδραση από εδώ και πέρα μεταξύ βουλευτών, ευρωβουλευτών, θεσμικών οργάνων και των τοπικών κοινωνιών από τις οποίες προέρχεστε εσείς, που εκπροσωπείτε εσείς εδώ. Είτε πρόκειται για ομολογιακές είτε για μη ομολογιακές οργανώσεις. Και νομίζω ότι υπάρχουν ε, δύο πεδία τομείς όπου μπορούμε να συνεργαστούμε. Πρώτον, στους επίσημους και τυπικούς τομείς πολιτικής που εντάσσονται σε αυτόν τον κοινωνικό πυλώνα που αφορούν την κοινωνική προστασία και φροντίδα, την προστασία των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, την προστασία των αστέγων και αυτή είναι τομείς δράσης και των θρησκειών και των εκκλησιών που πολλές φορές έρχονται και καλύπτουν τα κενά των κρατικών, των δημόσιων, των τοπικών ε, δημοτικών αρχών, γιατί όπως υπόθηκε και νωρίτερα, η οικονομική κρίση έπληξε σοβαρότατα ε, τις κοινωνικές δαπάνες και προκάλεσε μεγάλες κοινωνικές περικοπές. Το δεύτερο πεδίο συνεργασίας μας ε, έχει ευρύτερη, ε, ευρύτερο χαρακτήρα και ε, αφορά την ευαισθητοποίηση του κοινού για το γεγονός ότι η ολοένα και μεγαλύτερη ε, επέκταση μορφών ανταγωνιστικότητας ε, που οδηγούν σε, σε υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων ακόμα και σε σύγχρονη σκλαβιά απαιτεί την ανταπόκριση, την απάντηση της κοινωνίας η οποία θα πρέπει να επιμένει σε αυτά που υπόθηκαν στο προηγούμενο πάνελ. Εξασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ανάγκη να, καταστεί, να καταστούν υποχρεωτικά συγκεκριμένα πρότυπα και προδιαγραφές ανθρώπινης συμπεριφοράς, ανθρώπινης αξιοπρέπειας που δεν μπορούν να υπόκεινται στη λογική της ιδιωτικής οικονομίας και της αγοράς. Και το είπε και ο, ε, πρόεδρος του προηγούμενου πάνελ για τον Πρωθυπουργό που επισκέφθηκε το Στρασβούργο, την Ολμέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο πριν από δύο εβδομάδες, ε, ο οποίος υπερασπίστηκε την αγορά ως κινητήρια δύναμη και ως εργαλείο για την επίτευξη της επιθυμητής ανάπτυξης. Και όταν ρωτήθηκε για την κοινωνική διάσταση αυτής της οικονομικής ανάπτυξης, απάντησε ότι αυτό είναι αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους ξεχωριστά και ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το όραμα αυτό είναι βαθύτατα προβληματικό, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα και κύρια αποτελεί μια κοινότητα λαών. Δεν θέλω να ε, συνεχίσω και να καταχραστώ άλλο τον χρόνο. Και γι' αυτό και θα ολοκληρώσω με το τρίτο σημείο που θέλω να πω. Ο κατάλογος των συμμετοχόντων της σημερινής μας συνάντησης είναι πραγματικά πολλά υποσχόμενος. Από την άποψη ότι είναι ε, εξαιρετική η πολυμορφία των συμμετεχόντων στη σημερινή μας συνεδρίαση. Εγώ, ξέρετε, συμμετέχω σε πάρα πολλές συνεδριάσεις, σε καθημερινό σχεδόν επίπεδο, αλλά πρέπει να σας πω ότι σήμερα είστε πραγματικά... Ε, Υπάρχει μια εξαιρετική πολυμορφία σήμερα στους συμμετέχοντες σε αυτή τη συνεδρίαση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τονίζονται σήμερα αυτά, αυτή, τα κοινωνικά ζητήματα και θα μας βοηθήσετε με την συμβολή σας και τη συνεισφορά σας στη συζήτηση να μπορέσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά, από το δικό μας μετερίζει, να διαμορφώσουμε τον κοινωνικό πυλώνα με τέτοιον τρόπο και τις πολιτικές αυτού, ώστε να αποφέρουμε και να επιτύχουμε τα μεγαλύτερα δυνατά ε, αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Λοιπόν, θα σα παρουσιάσω τώρα του ομιλητέ μα. Δεν θα μπω όμω σε πολλά βιογραφικά στοιχεία για αυτού, ούτε τι ημερομηνίε γέννησή του θα σα πω. Έχουμε μαζί μα τον ε, δεσιμότητα Ντανιέλ Τοπάλσκι, που είναι έφορο τη της ε, Εκκλησία των Μεθοδιστών, υπεύθυνο, υπεύθυνο για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε μαζί μα τον Ρικάρδο Ντισένι, που είναι αρχιραβίνο τη Ρώμης από το 2001 και έχουμε και την Επίτροπο Birgit Μπρέκε Κλίφτον, ε, Επίτροπο της, ε, ε, του, του, της του στρατού της σωτηρίας. Κύριε έχει έχετε λόγο. Κύριε Αντιπρόεδρε, Μακίνες, κυρίες και κύριοι, Ευχαριστώ πολύ στα προφητικά λόγια του Ζακ που ήδη ο ε, Σεβασμιότατος Ιγνάτιος ε, ανέφερε ότι ε, δεν θα πραγματώσουμε με το όρομα για την Ευρώπη βασιζόμενοι αποκλειστικά και μόνο στην νομική πραγματοσύνη, αλλά χρειαζόμαστε να δόμαστε και ε, ψυχή στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Όλες οι αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ευρώπη η ειρήνη, λεγική ισότητα, ενότητα στην πυκλομορφία, δημοκρατία, δικαιοσύνη, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία και οικολογική βιωσιμότητα μπορούν να θεωρηθούν ως τμήμα της ε, ευρωπαϊκής ψυχής ενώ ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Πολύνος Πυλώνας μπορεί να αποτελέσει ένα τμήμα αυτής της ψυχής και ως ένα σημείο υπενθύμησης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε κοινέ αξίες και μεταξύ αυτών των αξιών βρίσκονται και οι αξίες ε, των ίσων ευκαιριών, της πρόσβασης στην αγορά εργασία, των δίκαιων ε, σχέσεων και συνδικών εργασία και τη κοινωνική προστασία και ένταξη. Η ευρωπαϊκή κοινωνία δεν μπορεί να μοιαστεί και να ε, συμπεριλάβει όλα τα μέλη της αν η Ευρώπη προσπαθεί μόνο να ε, επιτύχει την ενότητά της μέσω νομικών και οικονομικών μέτρων. Σήμερα βλέπουμε ότι η Ευρώπη ε, δυστυχώς ολοένα και, στην Ευρώπη ολοένα και αποδυναμώνονται αυτές οι βασικές της αξίες. Χρειάζεται όμως να γίνει και μια αναζήτηση ταυτότητας και κοινωνικών σχέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη ως Ήπειρος χρειάζεται για άλλη μια φορά να δώσουν μια συγκεκριμένη και σαφή εξήγηση για το ποιε είναι οι ρίζες της και είναι, ποιοι είναι οι στόχοι της. Και γι' αυτό νομίζω ότι ε, η διαδικασία του άρθρου 17 είναι πραγματικά απαραίτητη. Και αν ο διάλογος είναι πραγματικά ανοιχτός, διαφανής και τακτικός και αν ε, το, το, πράγματι ο καθένας προσέρχεται στο διάλογο αυτό όχι μόνο για να τοποθετηθεί αλλά και για να ακούσει τα αποτελέσματα μπορούν να είναι πολύ ενθαρρυντικά. Οι εκκλησίε μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν ε, στην κοινωνία μέσω του διακονικού τους έργου και μέσω από αυτήν την ε, διαδικασία εμείς προσπαθούμε πραγματικά μέσα από τη διακονία να προσφέρουμε τη συμβολή μας και μεταξύ των ανθρώπων στους οποίους φτάνουμε είναι άνθρωποι που έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω της φίλης του φίλου, της πίστης, ε, των, ε, της σωματικής του ικανότητας ή της ηλικία. Γιατί τα κάνουμε όλα αυτά και γιατί θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο στοιχείο της δουλειά μας. Γιατί πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ενώπιον του Θεού και ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι κατ' εικόνα του Θεού. Κάποιος μπορεί να πει ότι αυτό είναι ένα από τα βασικό, βασικά μας χαρακτηριστικά ως χριστιανικής διακονίας σε σύγκριση με τις κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν άλλες οργανώσεις και ιδιαίτερα οι μη θρησκευτικέ οργανώσεις. Αλλά όπως και να έχει γνωρίζουμε ότι η χριστιανική διακονία προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες σε όλους χωρίς αποκλεισμούς. Όπως γνωρίζετε, τα κράτη-μέλη έχουν ε, ελεύθερο το πεδίο όσον αφορά την εφαρμογή της, ε, αυτού του κοινωνικού πυλώνα και να πόκειται σε εκείνους για το κατά πόσο θα εμπλέξουν τι θρησκευτικέ οργανώσεις στη διαδικασία αυτή της εφαρμογής του κοινωνικού πυλώνα. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίω ότι οι εκκλησίε θα σταματήσουν το διακονικό τους έργο αν τα κράτη-μέλη αποφασίσουν ότι δεν θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της εφαρμογής του κοινωνικού πυλώνα ή θρησκευτικέ οργανώσει. Αντιθέτω, εμεί είμαστε πάντοτε ανοιχτοί να προσφέρουμε να δώσουμε από την πλευρά μας, να φροντίσουμε τους ανθρώπους μας, εκείνους που χρειάζονται ιδίως προστασία και υποστήριξη. Η Ενωμένη Εκκλησία των Μεθοδιστών είναι μια παγκόσμια εκκλησία η οποία διεξάγει το διακονικό της έργο σύμφωνα με, τους, με κοινωνικές αξίες που σε πολύ μεγάλο βαθμό ταυτίζονται με τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Προσπαθούμε πάντοτε να διαμορφώσουμε μια, ένα ήθος ε, θρησκευτικών κοινοτήτων σύμφωνα με αυτές τις κοινωνικές ε, αξίες και αρχές που θα οδηγήσουν βεβαίως σε μια δημιουργία μια μιας παγκόσμιας κοινωνίας η οποία αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές προκλήσεις. Στην Ευρώπη πολλές φορές τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Κάποιε φορέ οι κυβερνήσει προσπαθούν και οι δημόσιε αρχέ προσπαθούν να τηρήσουν αρχέ, την απόσταση από τι ε, θρησκευτικές οργανώσεις. Σε κάποιες πρώην κομμουνιστικές χώρες οι θρησκευτικέ οργανώσει ακόμα συνοδεύονται από επιφυλακτικότητα ω προς τη, στάση ε, των δημόσιων αρχών. Υπάρχει μια δυσπιστία ως προς τις ε, προθέσεις τους. Υπάρχει και μια ε, επικίνδυνη τάση σε αυτές τις χώρες να εθνικοποιηθούν οι ε, θρησκευτικοί θεσμοί και να μετατραπούν σε δημόσιους φορούς. Συνήθως ο, ο λόγος που προβάλλεται ή η πρόφαση αν θέλετε που προβάλλεται είναι λόγοι εθνικής ασφάλειας. Εμείς όμως εκφράζουμε βαθύτατη ανησυχία για τον περιορισμό των ε, θρησκευτικών δικαιωμάτων και της ε, ανεξιθρησκείας. Ένα σημαντικό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας που σας, που περιγράφω είναι πρόσφατες τροπολογίες σε βουλγαρικό, στο βουλγαρικό νόμο περί θρησκειών που μάλιστα ε, έλαβε, ε, ε, έτυχε ευρύτατη της κοινοβουλευτικής υποστήριξης και που δυσκολεύει πολύ την ε, δραστηριότητα των εκκλησιαστικών οργανώσεων στη χώρα αυτή. Ελπίζω λοιπόν ο διάλογος που διεξάγεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις θρησκευτικέ οργανώσεις να αποτελέσει ένα θετικό παράδειγμα το οποίο θα μιμηθούν και τα κράτη-μέλη. Ιδίως εκείνα στα οποία εντοπίζονται αυτές οι πολύ ανησυχητικές τάσεις που μόλις περιέγραψα. Μέσω του διαλόγου μπορούμε να οικοδομήσουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη ε, και έτσι να ανταποκριθούμε και στην κοινωνική αποστολή των οργανώσεων μας που δεν αφορά βεβαίως μόνο τις ε, χρηματοδοτικές πηγές ή τους πόρους που βεβαίως και μπορούν να μας βοηθήσουν, αλλά μπορούμε εμείς να προσφέρουμε εκτός από αυτά και εμπειρία, ανθρώπινους πόρους, αλλά και οργανωτικές ικανότητες στην παροχή αυτών των πολύ σημαντικών για την κοινωνία υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Reverend. Ευχαριστώ πολύ, δεσμότατε. Παρακαλώ τώρα τον Ραβίνο Ντισένι να λάβει το λόγο. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους οργανωτές αυτής της ε, διάσκεψης για την πρόσκληση και να πω ότι σε μια εποχή κατά την οποία μιλούμε για θρησκείες μόνο από την έποψη της αντιπαράθεσης μεταξύ πολιτισμών ή κοινωνικών ε, διεκδικήσεων η αλλαγή προοπτικής που προσφέρει η δική σας διάσκεψη έχει ουσιώδη σημασία Ιδιαίτερα λοιπόν το πρώτο ζήτημα πρέπει να διευκρινίσουμε, αλλά νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε και από τις προηγούμενες ομιλίες, είναι αν υπάρχουν αυτοί οι στόχοι ε, υπάρχει βέβαια ο κοινό στόχο οπωσδήποτε τη κοινωνική Ευρώπη, αλλά με ποιο τρόπο. Και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όσον αφορά τι εβραϊκέ κοινότητε, η κοινωνία στόχων δεν έχει να κάνει με την ανάγκη ή με κάποιους καιροσκοπικού, κάποιες καιροσκοπικές επιλογές και τη πρέπει να τονίσω ότι ένα αγαθό κοινό δεν μπορεί να θεωρηθεί δευτερεύον στόχος. Αλλά γιατί, γιατί αυτές οι αρχές, αυτές οι αξίες είναι κομμάτι της ε, κουλτούρας του πολιτισμού, των παραδόσεών μας. Έτσι λοιπόν ε, μιλούμε για την εργασία ως ε, στοιχείο εγγενές της θρησκείας και των αξιών μας στον Εβραϊσμό. Από τις απαρχές έχουν προαχθεί αυτές οι αρχές, τις έχει εκφράσει και στα λόγια των προφητών ε, η βίβλος και με τους νόμους μας. Η παραδόση λοιπόν Ιουδαϊκή μας λέει ότι η προστασία των πιο αδυνάτων είναι υποχρέωση. Πρέπει να πω ότι η εβραϊκή θρησκεία κυρίως ομιλεί, η εβραϊκή νομική ομιλεί κυρίως σε όρους υποχρέωσης και όχι ε, δικαιώματος. Βλέπουμε λοιπόν ε, στα τα βιβλικά ίχνη, βλέπουμε στο Ταλμούδ, βλέπουμε στο Λεβιτικό, στο Δευτερονόμιο. Ε, αναφέρονται ιδιαίτερα στο Ταλμούδ η σχέση μεταξύ επιχειρηματιών, εργαζομένων, μισθωτών, συμπεριλαμβανομένων και των διερμηνέων, λέει ο Ραβίνος. Ε, με προτάσεις που μπορούν να λύσουν ζητήματα ισορροπίας δυνάμεων και να αποτελέσουν έτσι ένα μοντέλο, ένα καλό μοντέλο για να επιληθούν τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Η της παράδοσής μας είναι το Σαμπάτ, το Σάββατο, με την απόλυτη υποχρέωση για ανάπαυση που ισχύει για όλους και που είναι η αρχή της εβδομάδας. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτούς τους, αυτές τις κοινέ αρχές και τις προτάσεις που μπορεί να προέρχονται από ένα πολιτισμό, μια κουλτούρα πανάρχια, αλλά ταυτόχρονα έχουν μεγάλη επικαιρότητα και μπορούν να, δίνουν να δώσουν πρωτότυπες λύσεις. Έχουμε ε, βάσει αυτό λοιπόν τη δυνατότητα να σκεφτούμε διάφορες διαφορετικές λύσεις. Πώς μπορούμε αυτό το, το εργαλείο, το μέσο να το εκφράσουμε σε όρους πραγματικούς. Θα μπορούσα να δώσω διάφορες ε, προοπτικές. Καταρχάς, πολύ σημαντικό είναι η μαρτυρία των αξιών, πολύ σημαντική για κάθε θρησκευτική αξία, η οποία δεν είναι ενότητα μόνο λόγω της θρησκεία ή λόγω των θρησκευτικών, ε, οικογενειακών ή άλλων δεσμών. Πρέπει να αποτελεί μαρτυρία ιδεών και αρχών. Και έτσι εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι κάποιες αρχέ ε, συνιστούν το ε, DNA μας, την ταυτότητά μας την πολιτιστική. Και πρέπει μια κοινότητα να είναι σε θέση να υπολογίζει στο γεγονό ότι υπερασπιζόμενοι αυτέ τι αξίε, προάγοντα αυτέ τι αξίε, θα έχει όλες ε, θα έχει την παρουσία της, θα είναι ολόκληρη. Δεν ε, ε, μιλώ μόνο για τα θέματα του ρατσισμού και της αδιαλαξίας, αλλά ακόμα και για τους ευρωπαϊκούς αυτούς κοινωνικούς, για πυλώνες. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η υποχρέωση της εκπαίδευσης, της πέδευσης για ολόκληρη την κοινότητα με στόχο την εξασφάλιση ελευθερίας και της ευημερίας της θρησκευτική ομάδας όχι μόνο γενικά που είναι πολύ σημαντικό βέβαια επειδή υπάρχει κάποιο δικαίωμα να είναι κανείς διαφορετικός αλλά γιατί και ταυτόχρονα έτσι προάγονται και προβάλλονται οι κοινέ αξίες. Η μαρτυρία λοιπόν και η εκπαίδευση είναι ζητήματα που θα συστήσουμε και πάλι. Αντίθετα από τις άλλες ε, μεγάλες ε, ε, ομάδες της θρησκευτικέ δεν έχει μετατραπεί σε, και θα το συζητήσουμε αυτό αν θέλετε, δεν έχει εκφραστεί σε κομματικούς όρους η εβραϊκή κοινότητα για διάφορους λόγους και αυτή πολύ σημαντική αν θέλετε μπορούμε πάλι να τους ε, συζητήσουμε πέραν της εξαιρέσεως του Μπούντ και αυτό είναι μια άλλη ιστορία ε, αλλά πάντως έχουμε πολύ σημαντικές προσωπικότητες που έχουν τις ρίζες του στην εβραϊκή θρησκεία και ένα όνομα που δεν χρειάζεται να σας συστήσω είναι αυτό της Σιμών Βέιλ και που με συνειδητό ή ασυνείδητο τρόπο και λόγω και της ιστορίας ε, που αντιμετώπισαν, που βρέθηκαν να ζουν, ε, αν, ανέλαβαν ένα καθήκον, επιφορτίστηκαν με ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό καθήκον. Αυτό που έλεγαν νωρίτερα, την εκπαίδευση που είναι το εβραϊκό DNA και που είναι απαραίτητη αρχή. Από το μεμονωμένο πρόσωπο τώρα στην παρουσία μέσα σε μια κοινότητα, το πρόβλημα είναι πολύ πιο περίπλοκο και απαιτεί από τις δύο πλευρές, δηλαδή κοινότητες θρησκευτικές αλλά και το κράτος μια προσπάθεια. Και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο εξαρτάται από μια αντικειμενική κατάσταση κινδύνου, μπορεί να είναι πραγματική ή ε, να θεωρείται ότι μπορεί να υπάρχει μια απειλή ως προς την ασφάλεια λόγω αντισημιτισμού, λόγω απειλών στην θρησκευτική ελευθερία. Εν πάση περιπτώσει είναι πολλές οι, πολλοί αγώνες ε, που έχουμε αντιμετωπίσει διάφορες αρχές και δομές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου μας έχουν βοηθήσει τακτικά. Η ελευθερία λοιπόν θρησκευτική θα έπρεπε να μπορεί κανείς να ανοίξει περισσότερο, να επιτρέπει να ανοίξει κανείς περισσότερο τα φτερά του και τις προοπτικές του. Μα θα μου πει κανείς, μα πρέπει κανείς να διαλέξει ένα κόμμα, μία πλευρά. Τη μία πλευρά ή την άλλη. Η θρησκευτική κοινότητα όμως είπα νωρίτερα ότι πρέπει να είναι έξω από τις κομματικές επιλογές. Και αυτό είναι το δύσκολο δύσκολη επιλογή. Και μια τελευταία σκέψη με κάποιες συγκεκριμένε ε, προτάσεις. Κάποια στιγμή και χωρίς, κάποια εποχή και χωρίς παρέμβαση κρατική, οι θρησκευτικές κοινότητες ήταν ε, εκείνες οι οποίες πάντοτε προσέφεραν όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Το άλλο το έχουμε δει με την ιστορία των νοσοκομείων που ε, εξασφάλιζαν την περίθαλψη και όπου εξασφάλισαν την περίθαλψη οι εκκλησίες, τώρα έχουν ε, μείνει ορισμένα μόνο που ανήκουν σε θρησκευτικέ κοινότητε. Έτσι λοιπόν οι θρησκευτικέ κοινότητε μπαίνουν μέσα σε συγκεκριμένα κομμάτια ε, που καλύπτουν ανάγκες της κοινωνίας πολύ περιορισμένα, ίσως όχι όμως περιθωριακά. περιθωριακά. Έχουμε ήδη παράδειγμα μια, ε, μια οργάνωση που λέγεται Χάτσολο, η οποία έχει ξεκινήσει από τις ΗΠΑ, έχει επεκταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και προσφέρει ε, περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ε, ανάγκης κατεπήγοντος περιστατικού. Υπάρχουν πολλές άλλες τέτοιες περιπτώσεις και γι' αυτό πρέπει να τονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο η θρησκευτική κοινότητα μπορεί και να αρχίσει με βάση τις αρχές να εντοπίζει το πρόβλημα, να προγραμματίσει, να οργανώσει, να διαχειριστεί τουλάχιστον βράχει και μέσο πρόθεσμα του σπόρους για την αντιμετώπιση του προβλήματο και πάντως μπορεί να αποτελέσει τον παράγοντα, τον φορέα τη αλληλεγγύη τη κοινωνική με αποτελεσματική δράση που θα διαφυλάξει την κοινωνία στην ενότητα αλλά και στις διαφορές της. όλα αυτά με δεδομένη τη δύσκολη εποχή που ζούμε μετά το 2001 που ξανά έφερε στο προσκήνιο παλαιές ε, διαφωνίες ή προκαταλήψεις. Ευχαριστούμε πολύ, Ραβίνα Ντισέιν. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Επιτρόπο Μπρίκε Κλίφτ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να συμμετάσχω στο διάλογο αυτό. Χαιρετίζουμε και εμείς αυτή την διαβούλευση και την αναγνώριση από την πλευρά των θεσμικών οργάνων ότι έχουμε κι εμείς ε, λόγο στη διαδικασία αυτή. Εγώ εκπροσωπώ το στρατό της σωτηρίας που ε, ιδρύθηκε πριν από 150 χρόνια στο πληττώνομενο από τη φτώχεια Ανατολικό Λονδίνο και έκτοτε ε, κηρύσουμε τον Ιησού Χριστό και την αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων χωρίς διακρίσεις. Και πλέον έχουμε παρουσία σε 130 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα τελευταία 40 χρόνια ε, εργάζομαι για τον στρατό της σωτηρίας και έχω ζήσει σε κάποιες από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο. Μεταξύ αυτών ε, και στο Πακιστάν και στο Μπαγκλαντέ. Έχω εργαστεί σε μια σειρά σλάμς ε, σε, σε παραγκουπόλεις, σε φτωχότατες περιοχές, αλλά έχω ζήσει και εργαστεί και σε πολύ φτωχές ε, περιοχές στην Ευρώπη. Πριν από κάποια χρόνια ε, επισκέφτηκα την Σλοβακία και εκεί επισκέφτηκα καταβλισμό Ρωμά και μπροστά μου αυτή τη στιγμή ε, έχω στο νου μου το πρόσωπο μιας μικρής, ενός μικρού κοριτσιού Ρωμά που είχε πάρα πάρα πολλές μέρες, ίσως και εβδομάδες να κάνει μπάνιο. Τα χεράκια της ήταν πάρα πολύ βρώμικα, ζούσε πραγματικά σε μια παραγκούπολη, χωρίς ε, στοιχειώδεις ε, εγκαταστάσεις προσωπικής υγιεινής ε, και μου φάνηκε ότι πραγματικά η ζωή της, από τη ζωή της έλειπε κάθε ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Διαβάζοντας όμως τα έγγραφα που είχαμε στη διάθεσή μας ε, πριν από τη σημερινή συνεδρίαση, αναρωτήθηκα θα έχει τελικά εκείνο το κοριτσάκι που συνάντησα στη Σλοβακία ένα μέλλον. Ζώντας πλέον σε ευρωπαϊκή χώρα, ο κοινωνικός πυλώνας πραγματικά θα φτάσει και σε εκείνη θα αλλάξει τις συνθήκες διαβίωσης της. Το ελπίζουμε όλοι μας φαντάζομαι, όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την αίθουσα. Και ε, το γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, του Στρατού της ε, Σωτηρίας συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις για την κατάρτιση αυτού του κοινωνικού πυλώνα. Συμμετείχαμε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, σε πάρα πολλές συνεδριάσεις από τότε που ξεκίνησαν οι διαβουλεύσεις που αφορούσαν την ε, συμπερίληψη των ανθρώπων με αναπηρίες σε υπηρεσίες στέγασης, ιατροφαρμακευτικής περιθέλευσης και προστασίας των αστέγων και ως φορέας κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής δράσης και με κινητήριο δύναμη τη χριστιανική μας πίστη ο στρατός της σωτηρίας έχει μεγάλη εμπειρία, μακρόχρονη εμπειρία με ανθρώπους που υφίστανται εκμετάλλευση, που απειλούνται από τη φτώχεια ή που ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά και στα 27 ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό υποστηρίζουμε αμέριστα τον ε, πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς θεωρούμε ότι έπαναπροσανατολίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη σε αυτά τα ζητήματα. Η αναγνώριση του κοινωνικού πυλώνα μέσω ενός πανευρωπαϊκού εγγράφου που εξασφαλίζει τα κοινωνικά πρότυπα και τι κοινωνικέ προδιαγραφέ σε ολόκληρη την Ευρώπη θα αποτελέσει εργαλείο στην υποστήριξη και την ενίσχυση τη κοινωνική ε, δικαιοσύνη, αλλά και στον ρόλο μα ω ε, παρόχου κοινωνικών υπηρεσιών και φροντίδα. Αναγνωρίζουμε λοιπόν την ανάγκη να υπάρξει σύγκληση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα για να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη ιδίω στι φτωχότερε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ανυψωθούν στο επίπεδο κοινωνική προστασία και κοινωνικών δικαιωμάτων που ισχύουν στις πιο αναπτυγμένες χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωση. και χαιρόμαστε πολύ που έχουμε να κάνουμε μια Ευρώπη η οποία τονίζει αυτή την ανάγκη της κοινωνικής ε, διάσταση και που υπερβαίνει ε, την ε, στενότητα των οικονομικών κριτήριων και τη οικονομικής διάσταση. Τρίτον, η αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή αυτού του κοινωνικού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και οι αρχές που κατοχυρώνονται στα άρθρα αυτού θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε σχέση με τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Εμείς λοιπόν ως στρατός της σωτηρίας υποστηρίζουμε φιλόδοξους στόχους ώστε να ενταχθούν και να συμπεριληφθούν τα κοινωνικά ζητήματα και να χρηματοδοτηθούν από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Οι αρχές του κοινωνικού ε, πυλώνα ε, απευθύνονται κυρίως σε εκείνους που έχουν ε, νόμιμη διαμονή, που βρίσκονται υπό καθεστώς ομαλότητας δηλαδή. Δυστυχώς όμως μένουν απ' έξω άνθρωποι που διαμένουν παράτυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι για παράδειγμα οι αιτούντες άσυλο. Αυτοί δεν προστατεύονται από τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον πυλώνα. Κατά τη γνώμη μας, πολύ συχνά, υπερβολικά συχνά, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγνοούν τα δικαιώματα, τις ανάγκες των αιτούντων άσυλο. Αυτοί οι άνθρωποι βεβαίω καλύπτονται από την Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και γι' αυτό λόγο έχουν δικαίωμα πρόσβαση σε ιατροφαρμική περίθαλψη, στέγαση, εκπαίδευση και εγκαταστάσεις υγιεινής. Ωστόσο, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις πολλές φορές αντιμετωπίζουν εμπόδια ως προς την παροχή τέτοιων κοινωνικών υπηρεσιών λόγω της, ε, της, της ε, πίεσης που ασκούν οι λαϊκιστές και οι εξτρεμιστικές φωνές που βρίσκονται σε άνοδο τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα άρθρα 11 και 17 της συνθήκης που αφορούν την κοινωνικοστική προστασία των παιδιών και των πλέον ευάλωτων ε, πληθυσμιακών ομάδων ισχύουν όμως και για τους ετούντε άσυλο, ενώ δυστυχώς ο κοινωνικός πυλώνας δεν κάνει ρητή αναφορά στη συμπερίληψη και αυτών των πληθυσμιακών ομάδων. Εμείς, ο στρατός της σωτηρίας, έχουμε θέση ως καθήκον και αποστολή μας την φροντίδα και αυτών των ανθρώπων. Όπου υπάρχει ανάγκη, εμείς βοηθάμε. Ανεξάρτητα από το αν κάτι τέτοιο κατεχειρώνεται σε ένα νομικό έγγραφο. Επιβεβαιώνουμε λοιπόν ότι οι υπηρεσίες που αφορούν την ανακούφιση της φτώχειας πρέπει να είναι ανοιχτές και προς τους ε, ε, ετούντες άσυλο, τους πρόσφυγες χωρίς χαρτιά και ότι και αυτοί αξίζουν τις προστασίες από την εκμετάλλευση. Για όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι πολύ θετική, ε, θετικό βήμα το κείμενο του κοινωνικού πυλώνα θεωρούμε ότι αποτελεί σοβαρότατη έλλειψη το γεγονός ότι δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν καλύπτονται από το κείμενο αυτό οι πρόσφυγες και τα άτομα χωρίς χαρτιά. Έχουμε ε, και κάποιες σκέψεις σε σχέση με το πεδίο και το εύρος των διαβουλεύσεων που προηγήθηκαν το κοινωνικό βαθμολόγιο που καταρτίστηκε. Δυστυχώς, αν δεν ληφθούν υπόψη οι πληθυσμιακές ομάδες που ανέφερα, δεν θα αποφέρει ολοκληρωμένα αποτελέσματα, ούτε θα, θα μας βοηθήσει να σχηματίσουμε μια σφαιρική εικόνα. Καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς δείκτες για να καταγράφουν όλες τις τάσεις και όλες τις εξελίξεις το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις δεν λογοδετούν και για αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα και χάσμα. Γιατί ακριβώς η εικόνα που θα σχηματίσουμε από το βαθμολόγιο που καταρτίστηκε δεν θα είναι ολοκληρωμένη. Το, ε, η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών ένταξης είναι απαραίτητη και αυτό προκύπτει και από την επικάλυψη και την ταύτιση των αρχών ε, του κοινωνικού πυλώνα με τους, ε, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ως λοιπόν διεθνής οργάνωση που δραστηριοποιείται όπως είπα σε 130 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο ε, κάνουμε έκκληση να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και εναρμόνιση μεταξύ των στόχων του κοινωνικού πυλώνα και των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη που έχουν καταρτιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για την παρουσίαση. Μας έχουμε λιγότερα από 20 λεπτά. Σας καλώ να τα αξιοποιήσετε. Βλέπω έναν κύριο εκεί που θέλει το λόγο, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω σήμερα ελληνικά ε, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία της παρουσίας των ευγενικών μεταφραστών μας. Και θα αναφερθώ σύντομα σε τρία σημεία που μου δώσαν ε, αφορμή να σκεφτώ οι τοποθετήσεις και των δύο ε, τόσο σημαντικών πάνελς που είχαμε σήμερα. Ένα πρώτο σημείο είναι το ζήτημα της μηχανοποίησης στην αγορά εργασίας. Η μηχανοποίηση οδηγεί σε απώλεια θέσεων. Και αν θέλουμε ε, αξιοπρεπή, όπως και όλοι θέλουμε που είμαστε σε αυτή εδώ την αίθουσα, αξιοπρεπή διαβίωση και αξιοπρεπές συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους, αυτό πηγαίνει μαζί πλέον με τη διαβίου εκπαίδευση. Οπότε ε, το, ο κοινωνικός πυλώνας θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο να πηγαίνει χέρι-χέρι με την διαβίου εκπαίδευση προκειμένου να ε, εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στους ανθρώπους που αναγκάζονται να αλλάξουν εργασία κάτω από τις νέες κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνει η αυτοματοποιημένη εργασία. Δεύτερο ζήτημα. Όλοι ζητάμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Το αίτημα αυτό που είναι κατανοητό ακολουθείται από ένα άλλο ερώτημα. Τι θα τον κάνουμε αυτό τον ελεύθερο χρόνο. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα στην Ευρώπη νιώθουν άβολα εκτός του χρόνου εργασίας και είναι καθήκον όλων ημών των ανθρώπων της Εκκλησίας, των εκπροσώπων των θρησκειών και όλων έχουν, όσων έχουν μια φιλοσοφική θεώρηση για τη ζωή, να δώσουν θετικό νόημα στην ανθρώπινη ζωή, για να μάθουμε ότι μπορούμε να είμαστε δημιουργικοί και εκτός εργασίας. Και ένα τρίτο ζήτημα, επειδή όλοι καταλαβαίνουμε μέρα με την ημέρα, όλο και περισσότερο, ότι για να έχουμε ένα κοινό, καλό, ευρωπαϊκό μέλλον, χρειάζεται να δουλέψουμε από κοινού στις κοινέ ευρωπαϊκές αξίες, ο κοινωνικός πυλώνας θεωρούμε ε, Μιλώ εδώ ως σύμβουλος του Γραφείου της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θεωρούμε, ότι ο κοινωνικός πυλώνας, ο ευρωπαϊκός κοινωνικός πυλώνας πρέπει να έχει στο κέντρο την οικογένεια. Να δοθούν δηλαδή κίνητρα μητρότητας και πατρότητας ώστε να μπορούν τα νέα ζευγάρια ειδικά σήμερα με τις σύγχρονες στις συνθήκες ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης να μπορούν τα νέα ζευγάρια να χαρούν από κοινού μητρότητα και πατρότητα. Διότι η οικογένεια είναι ο θεσμός ο οποίος διασώζει τις κοινέ ευρωπαϊκές αξίες. Και αν θέλουμε κοινέ ευρωπαϊκές αξίες πρέπει να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή οικογένεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Βλέπω μια κυρία εκεί πίσω στην αίθουσα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Heather Roy από την οργάνωση στην οποία συνεργάζεται το έργο το διακονικό των εκκλησιών αλλά και οι οργανώσεις προσφοράς ε, φιλανθρωπικής βοήθειας των εκκλησιών. Ε, θα ήθελα να συμφωνήσω με τα λόγια που ακούστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακούσαμε για το ρόλο των εκκλησιών στην κοινωνία ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι κάνει. Ε, νομίζω ότι οι ομιλητές μας σήμερα κάπως το υπενήχθησαν. Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων είναι ένας στόχος και σημαίνει αξίες, 28 αξίες για αυτούς που ζουν στην Ευρώπη, τους πολίτες Ευρώπης, αλλά δεν είναι το τέλος, ε, μπορεί να είναι ένα μέσο για να φτάσουμε στο τριπλό α που φαίνεται να θέλει ο κύριος Γιουνκέρ να εξασφαλίσει ως αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και γι' αυτό θα έπρεπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνάουν σταματοφύλακα για τον τρόπο με τον οποίο σε εθνικό επίπεδο υλοποιείται αυτό ο κοινωνικό πυλώνα μου, γιατί μόνο εκεί θα μετρηθεί η επιτυχία ω προ τον κοινωνικό πυλώνα και ταυτόχρονα θα ήθελα το Κοινοβούλιο να προασπίζετε τον πυλώνα, να προασπίζετε κάθε υποβάθμιση των δικαιωμάτων και αξιών που ε, περιλαμβάνει ο κοινωνικό πυλώνα, ακόμα και αν πρόκειται για επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι πολύ σημαντικό όταν την, ε, του χρόνου θα συναντήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ίσω υπάρξει συζήτηση για κατάργηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και πρέπει το Κοινοβούλιο επίσης να αναπτύξει την δραστηριότητά του ως ε, σώματος νομοθετικού, ως σώματος χάραξης πολιτικής, γιατί έχουν γίνει ήδη προτάσεις για το συγκερασμό βίου ε, οικογενειακού και ε, επαγγελματικού, αλλά μια και με τη συναποφασία έχει αυτή την εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, θα θέλαμε να ενισχύσει τις προσπάθειες των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των εκκλησιών, των φιλανθρωπικών οργανώσεων που στηρίζονται στην πίστη και να συμπληρώσει το έργο τους. Και βέβαια η υλοποίηση του πυλώνα πώς θα προκύψει ε, μέσα από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οικονομικό σκέλος δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, βλέπω έναν κύριο εδώ και μετά η κυρία πίσω. Από το, τη Βρετανική εταιρεία ε, ε Ο αρχιραφήνος της Ρώμης μας έδωσε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της Χοτσόλα που προσφέρει υποστήριξη σε έκτακτες ανάγκες. Και οι υπηρεσίες αυτές βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό μάλιστα βρίσκεται, ε, η, τα, τα, τα κεντρικά γραφεία αυτών των ε, οργανώσεων ε, βρίσκονται στο Λονδίνο σε μια περιοχή όπου ζουν ε, πάρα πολλοί Εβραίοι. Πώς μπορούν λοιπόν οι μη θρησκευόμενοι άνθρωποι να συμβάλλουν σε μια τέτοια διαδικασία, πιστεύετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας καλέσω όλους να υποδεχθούμε, να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Ταγιάννη. που μόλις εισήλθε στην αίθουσα. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την ε, κυρία που της είχα υποσχεθεί ότι θα της έδινα το λόγο. Ο διάλογος συνεχίζεται. Αν θέλετε να ακούσετε και μια παρέμβαση, κύριε Πρόεδρε, και στη συνέχεια να λάβετε το λόγο, βεβαίως είναι και αυτό μια δυνατότητα. Ο Πρόεδρος λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ θερμά, αγαπητοί αντιπρόεδροι, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Για πολλά χρόνια, για δύο μισή χρόνια, είχα την ευθύνη του διαθρησκευτικού διαλόγου. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να λάβω μέρος σε αυτήν την ε, συνάντησή σας που οργάνωσε η Αντιπρόεδρος κυρία Μαγκίνες, στην οποία έχω παραδώσει τη σκητάλη θεωρώντας ότι θα ήταν και ικανότερη να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα. Καθήκοντα και λεπτά βέβαια, γιατί δεν τίθεται μόνο ζήτημα να εξασφαλιστεί μια συνάντηση των θρησκευτικών ηγετών που ούτως ή άλλως πάντα είναι διαθέσιμη στο διάλογο, γιατί από εκεί και πέρα έρχεται η ώρα της υλοποίησης της, στην πράξη του διαλόγου σε κάθε επίπεδο. Όταν μιλούμε για κοινωνικό πυλώνα και το ρόλο που μπορούν ε, οι θρησκείες να αναλάβουν, τα πράγματα περιπλέκονται κάπως, γιατί στο κόσμο της εργασίας, του σχολείου, με όλες τις εγγυήσεις για την προστασία που ζητούν ε, οι πολίτες στον κόσμο του διαλόγου, της καθημερινής ζωής, ε, της καθημερινότητας από τις θρησκείες τους, γιατί είναι εύκολο να λέει κανείς στο τραπέζι των ισχυρών συμφωνούμε, αλλά όταν έρθει η ώρα να βρεθούμε αντιμέτωποι με διαφορετικές ε, συνήθειες, παραδόσεις, κουλτούρες, οι θρησκευτικές επιλογές, τα πράγματα δυσκολεύουν και νομίζω ότι εδώ έχουμε το καλύτερο εργαλείο να ενισχύσουμε την αμοιβαία κατανόηση, την άλληλο κατανόηση. Αλλά και μια κοινωνική πολιτική. Η εργασία είναι αυτή που εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια στον άνδρα και τη γυναίκα. Η ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών όταν ορισμένοι δεν είναι σε θέση καν να περιγράψουν ποια μπορεί να, είναι ο ρόλος της ε, γυναίκα και θρησκευτικέ ε, αρχές ακόμη φαίνεται να μην μπορούν να ερμηνεύσουν τη θρησκεία ή την ερμηνεύουν προ μία κατεύθυνση μόνο. Έχουμε δει όμω εδώ και οι μουσουλμάνες γυναίκες να καταβάλουν προσπάθειε για συμμετοχή στη συζήτηση. Η θρησκευτική πτυχή πιστεύουμε μπορεί να βοηθήσει στην εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή. Μπορούν και οι θρησκευτικέ οργανώσεις να βοηθήσουν στην προετοιμασία για την ένταξη στην αγορά εργασία στην εργασία ε, γιατί βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη, στην ε, ιδιαίτερη ιδιαίτερα έχουν και σχολές ε, και επαγγελματικές και σχολές κατάρτισης ε, των εργαζομένων που οργανώνουν οι ίδιες. Και πάντα βέβαια υποστηρίξαμε την Ευρώπη που ευνοεί την ανάπτυξη και μειώνει τις αποστάσεις μεταξύ πλουσίων και φτωχών. 23 εκατομμύρια ε, στην Ευρώπη νέοι από τα 15 έως τα 23 κινδυνευ... δεν έχουν ούτε εκπαίδευση ούτε ε, απασχόληση. 130 ε, εκατομμύρια βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχεια. Είναι η πρώτη γενιά αυτή που μεγαλώνει τώρα που κινδυνεύει να έχει χειρότερε προοπτικέ από αυτέ των γονιών τη. Και για λόγους ηθικούς ακόμα πρέπει οι θρησκείες να κάνουν ό,τι μπορούν για να προσφέρουν ελπίδα στους νέους σε αυτούς που βρίσκονται σε πιο αδύναμη θέση. Σε αυτούς που έχουν ανάγκη αυτή την υποστήριξη. Βέβαια αναφέρομαι και στην ενσωμάτωση και των μεταναστών στο χώρο εργασίας, όλων αυτών που προέρχονται από διάφορα μέρη του κόσμου και μπορούν μέσα από μια θρησκευτική οργάνωση να βρουν ευκαιρίες ενσωμάτωσης, ενσωμάτωσης ένταξης στην κοινωνία. στην ε, πόλη μου και το γνωρίζει ο Ραβενό ε, Ντισένιο. Παραδείγματι, η Καθολική Εκκλησία έχει αποδεχθεί σε μια προσπάθεια για ενσωμάτωση των Φιλιππίνων, των Φιλιππινέζων, που είναι πολλοί, έρχονται από μια άλλη ήπειρο, πολλέ φορέ δεν γνωρίζουν καν τη γλώσσα, αλλά ήδη έχει μπορέσει η Εκκλησία, χάρη και σε ιερεί που έχει φέρει από τι ε, Φιλιππίνε και μιλούν τη γλώσσα τους, να τους ενσωματώσει στην κοινωνία. Το ίδιο και με προσπάθειες αντίστοιχε για ε, προσπάτης Ισλαμικής πίστεως. Η διευκόλυνση επίσης του κοινωνικού διαλόγου είναι μια άλλη συμβολή των θρησκειών. Είδαμε σήμερα στον Ιταλικό τύπο επί και μας κατέπληξε αυτό ότι γιατί έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις και με το Ραβίνο Ντισένιο, συναντήσεις μεταξύ καθολικών, Εβραίων και μουσουλμάνων για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, την ανάκτηση για την κοινωνία των ναρκωμανών. Είναι ένα θέμα επίσης πολύ σημαντικό στο οποίο μπορεί να συμβάλλουν οι εκκλησίες. Στο Κότεμπορκ υπογράφηκε μια συμφωνία. Όμως τα κοινωνικά προβλήματα είναι πολύ ευρύτερα από το σύνολο του καθενός μεμονωμένου προσώπου με τα προβλήματά του και τον αποκλεισμό της κοινωνίας. Κυρίως για τους νέους ή τα άτομα με αναπηρία ή πρόσβαση στην αγορά εργασίας, παράδειγμα, ότι μπορεί να διευκολυνθεί χάρη στις θρησκείες, στις σκεφτικές οργανώσεις από αυτή την έποψη. Επίσης έχουμε ασχοληθεί με την οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζομένους, με την νομοθεσία για το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης, το πρόγραμμα δράσης για την κάλυψη του, του, κενού, της διαφοράς, μεταξύ αμοιβ, για, της διαφοράς στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όλα αυτά για να μπορούμε να εργαζόμαστε μαζί. Και πιστεύω ότι και οι θρησκείες μπορούν να συμβάλλουν. Είμαι ακριβνής υποστηρικτής της επικουρικότητας και της εγκάρσιας αυτής, γιατί και οι θρησκείες μπορούν να προσφέρουν με το εξαιρετικό εργαλείο που έχουν της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συμπερίληψης που μπορούν να, που χάρη σε αυτό μπορούν να κάνουν εξαιρετική δουλειά, με την κατάρτιση, με την εκπαίδευση των νέων, γιατί αν δεν δώσουμε αξίες στα παιδιά μας, στους νέους μας, κινδυνεύουμε να έχουμε μια κοινωνία όλο και πιο κατακαιρματισμένη και αποψηλωμένη, έτσι ώστε θα φτάσουμε σε έναν κόσμο που δεν θα υπάρχουν πια υποχρεώσεις, όπου οι νέοι μας θα θεωρούν ότι έχουν μόνο δικαιώματα και, ότι, και θεωρώ ότι ίσως μόνο οι θρησκευτικοί παιδεία μπορεί να δώσει στα παιδιά μας αυτή την πτυχή, ε, το δίπτυχο αυτό, ε, υποχρέωση και δικαίωμα ότι είναι η του νομίσματος Και θα ήθελα, υπό αυτή την έποψη, να ζητήσω όλο και περισσότερη προσπάθεια ε, από τις θρησκευτικέ οργανώσεις, από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, ε, και έχω δώσει ήδη ένα στοιχείο το οποίο με ανησυχεί ιδιαίτερα σε σχέση με την πατρίδα μου την Ιταλία για την υποχώρηση της παρουσίας όλων των ε, ε θρησκειών. Είμαι πεπισμένος ότι οι θρησκείες έχουν θεμελιώδη ρόλο στη ζωή της, ε, του καθενός μας και μπορεί η θρησκεία να δώσει λύσεις και για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Οι θρησκείες στις θρησκευτικέ οργανώσεις δεν είναι με κυβερνητικέ οργανώσεις βέβαια. Έχουν διαφορετικά καθήκοντα. Ωστόσο η κατάρτιση των νέων, η παιδεία και οι αξίες που, προσφέρουμε στους, που προσφέρουν στους νέους είναι νομίζω το κύριο καθήκον τους σε μια κοινωνία όπου υπάρχουν ε, νέοι πιστοί. Μια κοινωνία που έχει νέους πιστούς είναι μια πιο πλούσια κοινωνία και μια κοινωνία που θα δουλέψει με πλούτο τους νέους, με κύριο πόρο τους νέους. Αυτό μπορούν να προσφέρουν οι μονοθεστικές οργανώσεις, ε, εκκλησίες, συγγνώμη, στους νέους μας και αυτή την κοινωνική συμπερίληψη. Και έτσι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί, όλοι μαζί στην Ευρώπη μπορούμε να συμβάλλουμε για την κοινωνική συμπερίληψη και τον κίνδυνο να χαθούν, να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο να χαθούν αυτές οι αξίες. Μια κοινωνία με αξίες μπορεί να ζήσει. Μια κοινωνία χωρίς αξίες κινδυνεύει να καταρρεύσει. Βεβαίως είναι πολύ σημαντική η εργασία ως κομμάτι της ζωής. δεν αφορά μόνο και αποκλειστικά τη ζωή μας. Είναι ένα μέρος της ζωής μας, όπως είναι ένα μέρος της ζωής μας, όπως διαπνέει όλη μας τη ζωή η θρησκεία. Και σε αυτό έχουν οι θρησκευτικέ ε, οργανώσεις και οι θρησκευτικοί ηγέτες το καθήκον να βοηθήσουν πάνω απ' όλα τους νέους για να ζήσουν σε μια Ευρώπη όπου δεν μετράει μόνο το χρήμα. Η γραφειοκρατία, οι δομές οι κρατικές, αλλά οι αξίες. Και στον χώρο της εργασίας είναι σημαντική η υποστήριξη. Αυτό που κάνουμε λοιπόν με το χώρο εργασίας που πρέπει να κάνουμε είναι να μην γίνει σημείο διχασμού ή στοιχείο διχασμού το θρησκευτικό στοιχείο, αλλά στοιχείο ένωσης. Όχι μίσους λοιπόν, αλλά ένωση και αγάπη. Χριστιανοί, Εβραίοι και Μουσουλμάνοι ζουν μαζί στην Ευρώπη. Ακολουθούν το πιστεύω τους τα θρησκευτικά αλλά δεν πρέπει κανείς να χρησιμοποιεί τον Θεό για να καλλιεργεί διχόνοιες. Θα ήταν πολύ κακό αυτό για τις κοινωνίες μας, θα ήταν ένα χείριστο παράδειγμα και μήνυμα για τους νέους μας. Ελπίζω αυτός ο διάλογος να φέρει θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία μας και ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο Μαγκίνες. που ανέπτυξε το συγκεκριμένο αυτό θέμα. του κοινωνικού διαλόγου, της κοινωνικής συμπερίληψης. Ένα διαλόγου που μπορεί να επιτρέψει να εξασφαλιστούν πιο φιλόδοξοι στόχοι. Ευχαριστώ την κυρία Μαγκίνες. Ολοκληρώνει το ρόλο της και υλοποιεί τα καθήκοντά της ως Αντιπροέδρου. Συνεχίζει λοιπόν το έργο που είχα εγώ πριν. Είμαστε σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό και δεν μπορώ παρά να υπερνέσω το έργο της. Σας ευχαριστώ θερμά. Ένα μήνυμα από του διερμηνεί. Ε, Δυστυχώ βρισκόμαστε στην 22η ημέρα των κινητοποιήσεων μα. Δυστυχώ η μερα των κινητοποιησεων μα δυστυχω η διοικηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει σκληρύνει μάλιστα τι τάσει αντί να υποχωρήσει. Και γι' αυτό σε ένδειξη διαμαρτυρία δυστυχώ η διερμηνία θα διακοπεί όπω προβλεπόταν από το πρόγραμμα. Become a guarantee for the implementation of the pillar. Because we were discussing what different uh, religious and non-religious uh, organizations could do to implement the pillar